Okay. So, welcome everybody. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους σε αυτή την συνεδρία της Επιτροπής μας. Καταρχήν θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω κανέναν να έχει αντίρρηση. Οπότε εγκρίνεται. Δυστυχώς όμως έχω κάποιες ανακοινώσεις του Προέδρου, ως συνήθως. Καταρχήν υπάρχει, πρόκειται για κοινή συνεδρίαση αύριο το απόγευμα με την Επιτροπή Απασχόλησης Οικονομικός Διάλογος με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών και Εργασίες Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κοινή συνεδρίαση ΕΚΟΝ και απασχόλησης από τις 3.30 μέχρι τις 5.30 στην 5G3 εδώ, σε αυτή την αίθουσα δηλαδή. 7 Νοεμβρίου έγινε τριμερής διάλογος ε, με την CRA 3 με τρίτες χώρες όπου έχουμε διάφορα κρεμή ζητήματα όπως ε, τα δάνεια, τα χρέη, ε, η κυκλική εναλλαγή. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να καταλήξουμε υπό την Κυπριακή Προεδρία στις 13 ε, Νοεμβρίου ξανά έχουμε συνάντηση με τον Επίτροπο Μπαρνιά για το διπλό πακέτο ε, το Τούπακ επόμενη συνεδρίαση προβλέπεται για τις 15 μια πρόοδος Όσον αφορά όμως ε, το υπερβολικό χρέος ε, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος. Έχουμε και κάποια σημαντικά θέματα πολιτικής, ε, πολιτικού χαρακτήρα, κυρίως το κεφάλαιο 3 της έκθεσης Φερέρα που προβλέπει το Ταμείο Διάσωσης και τις διατάξεις περί ανάπτυξης. Τώρα όσον αφορά την έκθεση Γκοζές υπάρχουν θέματα για τη φορολόγηση και τις ε, ψηφοφορίες, ε, αντίστροφη ειδική πλειοψηφία και σήμερα συνεχίζεται η συζήτηση για την ε, CRD4 Αυτέ ήταν οι ανακοινώσει μου και περνάω με τα χαρά στη τρίτο σημείο, ανταλλαγή απόψεων και οικονομικό διάλογο με τον Ισπανό Υπουργό Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας. Πρόκειται για την τρίτη επαφή με Υπουργό Οικονομικών Οικονομίας ε, ενός κράτους μέλους ε, σύμφωνα με τις διατάξεις προβλέπονται από το εξαπλό πακέτο, το Six Pack. Ε, έχουμε τη σειρά της Ισπανίας σήμερα. Οι συντονιστές της ΕΚΟΝ αποφάσισαν να καλέσουμε και την Ιταλία για τη σημερινή συνεδρία, αλλά δυστυχώ ο Ιταλό Υπουργό Οικονομία δεν μπορούσε να έρθει. η προσωπία ΕΚΟΝ ε, ανέφερε το θέμα ε, στον Ιταλό Υπουργό που συμφώνησε να έρθει στην ΕΚΟΝ πριν το τέλο του έτου. Οπότε προσβλέπουμε στον οικονομικό διάλογο με την Ιταλία. Επίσης, προς ενημέρωσή σας, να σας πω ότι οι συντονιστές αποφάσισαν να καλέσουν τους Υπουργούς Οικονομικών για Γαλλία και Γερμανία και με τα χαρά σας αναφέρω ότι και οι δύο αποφάσισαν, ε, μάλλον, απάντησαν μάλλον να έρθουν ε, και ο Μοσκοβίτση και ο Σόιμπλε, μάλλον στις 3 Δεκεμβρίου. θα σας έρθει επιβεβαίωση αργότερα. Και τώρα με τα χαρά μου θα δώσω το λόγο στον Ισπανό Υπουργό Οικονομίας, Έχετε γύρω στα 10 λεπτά και σίγουρα θα έχουμε πολλές ερωτήσεις για σας μετά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως Υπουργό Οικονομικών της Ισπανίας αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή εδώ που βρίσκομαι εδώ στην καρδιά της ε, Ευρωπαϊκής ε, Δημοκρατίας και να σας παρουσιάσω την οικονομική στρατηγική της Ισπανίας εν ώψη των ε, τεράστιων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Όπω όλοι γνωρίζετε είναι περίπλοκη κατάσταση Υπάρχει η παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση που επηρεάζει και τις ανεπτυγμένε και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Για την Ευρωζώνη, πέρα τη γενικευμένης επιβράδυνσης, έχουμε και ένα πρόβλημα βεβαιότητας, ε, αμφιβολίες για το ευρώ και κρίση εμπιστοσύνη ε, των διεθνών κεφαλαίων αγορών σε ό,τι αφορά την Ευρωζώνη. Είμαι πεπισμένο όμω ότι για να ξεπεράσουμε αυτή αυτή την κατάσταση και για να ενισχυθούμε θα πρέπει να επενδύσουμε σε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο για τη βελτίωση της διαφάνειας, της δημοκρατίας και της ε, ευθύνη και λογοδοσίας στη λήψη των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της. Γι' αυτό και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτοί οι οικονομικοί διάλογοι αποτελούν ένα θεμελιώδες στοιχείο και πολύ σημαντικό στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για να βελτιωθεί η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ιδιαίτερη χαρά θα έρθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσε φορέ χρειαστεί για να ενημερώσω του Ευρωπαίου πολίτε για το οικονομικό πρόγραμμα τη Ισπανία και την συνεισφορά μα σε μια οικονομική και νομική ένωση που θα είναι εύρωστη και ισχυρή. Θα σα εξηγήσω πρώτα τι μέτρα έλαβε η Ισπανία προσπαθώντας να αντιμετωπίσει αυτές τις αβεβαιότητες και τις ανασφάλειες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα για να βελτιώσουμε τις ανισορροπίες που σώρευσε η Ισπανική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Τους τελευταίους μήνες η Ισπανική κυβέρνηση θέτησε πακέτα μέτρων που κατά τη γνώμη μας είναι και θαραλέα και συνεκτικά και συνεπή. Δύο είναι οι βασικοί μας ε, στόχοι στην οικονομική πολιτική και αλληλένδετοι μάλιστα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε οικονομική ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης ε, και φυσικά να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι, επαναλαμβάνω, αλληλένδετοι οι δύο στόχοι. Στηριζόμαστε σε τρεις βασικούς άξονες ε, την μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα για να εξασφαλίσουμε ε, ρευστότητα κεφαλαίου, να διορθώσουμε τις τραπεζικές ανισορροπίες και να προσπαθήσουμε να ανακεφαλαιοποιήσουμε και να αναδιαρθρώσουμε τις τράπεζές μας. Δεύτερον, πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για να ενισχύσουμε το δυναμικό της οικονομικής ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας και επίσης ε, ακράδαντη υπεποίθηση να εξηγιάνουμε τα οικονομικά μας σε ό,τι αφορά το χρηματοπιστωτικό κλάδο, θα ήθελα να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του 2012 προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε μια διαφανή ισορροπία και επιδείξαμε τεράστια αξιοπιστία. Προσπαθούμε να θεωρήσουμε τις κεφαλαϊκές ανάγκες του, χρηματο... του τραπεζικού μας τομέα. Και μάλιστα αυτή η προσπάθεια έγινε για το 90% της τράπεζας και ιδιαίτερα για όλο το χαρτοφυλάκιο των πιστώσεων των οργανισμών αυτών. Και μετά τα stress test καταλήξαμε στα εξή συμπεράσματα. Το 70% του ισπανικού χρηματοπιστωτικού τομέα είναι υγιής, φερέγγιος και δεν χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση. Επίσης, το 90% των κεφαλαίων ε, στηρίζονται, συγκεντρώνονται σε τέσσερις ε, τράπεζες που ήδη ε, εθνικοποιήθηκαν. Και μάλιστα υπάρχει και ένας αρμόδιος οργανισμός για την αναδιάρθρωση του ισπανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Και μάλιστα πρόκειται για τράπεζες που είναι πάνω κάτω από το 20% του συνολικού τραπεζικού κλάδου της Ισπανίας. Ό,τι αφορά τις κεφαλαϊκές ανάγκες, έχουμε υπολογίσει ότι είναι γύρω στα 60 δις. Και ε, τελικά οι πραγματικές είναι κάτω από 40 δις, δηλαδή λιγότερο από 4% του ισπανικού ΕΠ. Πρόκειται για ένα ποσό πολύ χαμηλότερο από την γραμμή που, των 100 δις που εγκρίθηκε για την Ισπανία για, για την ενίσχυση. Καταρχήν θέλουμε μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού από τις τράπεζες στην, στο, στην κακή τράπεζα που θα διαχειρίζεται αυτά τα επισφαλή ενεργειακά, ε, ε, στοιχεία του ενεργητικού, αξιολόγηση των στοιχείων του ενεργητικού, κατανομή του βάρους όσο αφορά το χρέος και τα επιμέρους στοιχεία και επίσης προσπάθεια ανέβρεσης ιδιωτικού κεφαλαίου αντί για κρατικές βοήθειες και ενισχύσεις. Με αυτά τα αποτελέσματα συνεχίζουμε τη στρατηγική της Ισπανικής κυβέρνησης που υιοθετήσαμε στις αρχές του έτους με μέτρα για την βελτίωση τη της επάρκειας των πόρων των τραπεζών. Επίσης, στο μέλλον θα προβούμε σε ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που τη χρειάζονται και θα θέσουμε σε λειτουργία τη γνωστή ως κακή τράπεζα, που θα τεθεί σε λειτουργία από την 1η Δεκεμβρίου του τρέχοντο έτου, όπω προβλέπεται στο μνημόνιο συνεννόησης που συνυπογράψαμε με του εταίρους μα. Οπότε το Δεκέμβριο η προσπάθεια ρηξικέλευτη αναδιάρθρωση και εξηγίαση του τραπεζικού τομέα που ξεκίνησε το Φεβρουάριο θα έρθει σε πέρα. Έχουμε, ε, θα έχουμε ένα χρηματοπιστωτικό χάρτη με λιγότερε τράπεζε από 50 θα έχουμε σε 12 περίπου τέτοιες, τέτοιους φορείς, πολύ πιο φερέγγιους όμως και πλήρως ε, ε, ε, υγιείς. Όπως ανέφεραν η ΕΚΤ, η Κομισιόν και το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο, τηρούμε πιστά και με επιτυχία το, το, τη συμφωνία που έχουμε υπογράψει με τους εταίρους μας. Έχουμε ένα διαφανές πλέον πλαίσιο για την, υλοποίηση, για την αντιμετώπιση των τραπεζικών κρίσεων, μάλιστα πρωτοπόρο στην Ευρώπη. Και μάλιστα προλάβαμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συνδεδεμένη διαχείριση των προβληματικών τραπεζών και απαλλάσσοντας τους φορολογουμένους. Επίσης έχουμε και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις ε, προκειμένου να ενισχύσουμε το δυναμικό της ισπανικής οικονομίας, ε, κυρίως στον τομέα της προσφοράς. Μάλιστα, έχουμε υιοθετήσει ευρύτατε οικονομικέ μεταρρυθμίσει μέσω και μακροπρόθεσμα, προκειμένου να διορθώσουμε τι ανισορροπίε τη ισπανική οικονομία. Σε λιγότερο από 11 μήνε, καταλήξαμε σε ένα σημαντικό πακέτο διαρθρωτικών μέτρων. Καταρχήν, ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση τη αγορά εργασία, ε, κέρια για την Ισπανία, δεδομένων των απαράδεκτα υψηλών ποσοστών ενεργείας που μαστίζουν τη χώρα μου. Έχουμε τρία βασικά στοιχεία που πιστεύουμε ότι θα θέσουν πέρα στη ρεκαψία της αγοράς εργασίας. Καταρχήν προβλέπουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα στον τομέα των επιχειρήσεων ώστε να προσαρμόσουμε τη διαχείριση των πόρων στις οικονομικές συνθήκες. Επίσης, ε, οι επιχειρηματικές συμβάσεις θα υπηρεσχύουν των ε, τοπικών ή και επίσης λάβαμε πολύ σημαντικά μέτρα για την απελευθέρωση του τομέα των υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά το στεγαστικό κλάδο και ιδιαίτερα ε, στα ενίκια, έχουμε πια μεγαλύτερη ελαστικότητα και ασφάλεια δικαίου. Σε ό,τι αφορά το λιανεμπόριο, λιανικό εμπόριο, έχουμε άρση των διοικητικών φραγμών και άλλων φραγμών που εντοπίσαμε. Επίσης, ε, είχαμε μεταρρύθμιση της παιδείας και της δημόσιας υγείας. Όλα αυτά τα μέτρα ήδη φέρουν καρπούς, όπως είπα και προηγουμένως. Και πιστεύουμε ότι έτσι θα καταλήξουμε σε ένα νέο μεταρρυθμιστικό πακέτο. Έτσι η Ισπανία όχι μόνο τηρεί τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αλλά όπως αναγνώρισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ακόμη πιο φιλόδοξη ως προς αυτές τις συστάσεις. Ορισμένα από τα μέτρα είναι τα εξή. Καταρχήν, δημιουργία μιας ανεξάρτητης φορολογικής αρχής που θα ενισχύει την ε, αφαρμογή της, του νόμου της ε, φορολογικής δημοσιο, δημοσιονομικής δημοσιότητας. Ε, προσπαθούμε να θέσουμε τέρμα στον κατακαιρματισμό της εθνικής αγοράς. Βέβαια, θα έχουμε 1,5% αύξηση σχέση με το ΑΕΠ. Επίσης, απελευθέρωση κάποιων υπηρεσιών, ώστε να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό και βελτίωση των ενεργών πολιτικών απασχόλησης και κατάρτισης. Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Θα υιοθετήσουμε μέτρα για να προσαρμόσουμε την πραγματική ηλικία συντάξιμου με την νόμιμη ηλικία. Επίσης, προβλέπουμε κάποιες αναλλακτικές λύσεις για τη χρηματοδότηση χρηματοδότηση σχέση με την ε, τραπεζική χρηματοδότηση των ισπανικών επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, ανάπτυξη εναλλακτικών αρχών, ε, αγορών αξιών, καλύτερη διαχείριση του κινδύνου και βελτίωση του εθνικού συστήματο εγγυήσεων για να εγκριθούν οι χρηματοδοτήσει μέσω και μακροπρόθεσμες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τρίτο πυλώνας τη οικονομική πολιτική ε, τη ισπανική κυβέρνηση είναι φυσικά η αναζήτηση τη βιωσιμότητα μέσω πρόθεσμα των οικονομικών τη Ισπανία, ό,τι αφορά τη δημοσιονομική πολιτική. Θα μειώσουμε το δημοσιονομικό μα έλλειμμα σε πάνω από 2,5 ποσοστιαίε μονάδε, μάλιστα σε μια κατάσταση οικονομική ύφεση και με μείωση του ΑΕΠ που υπολογίζεται γύρω στο 1,5%. Θα ήθελα επίση να σας υπενθυμίσω τα σημαντικά μέτρα που εθέτει η Ισπανική κυβέρνηση για να μειώσει το έλλειμμά της τα επόμενα χρόνια. Καταρχήν ως προς τα έσοδα. Ε, συνολική προσπάθεια 40%. Έχουμε αύξηση του φόρου περιουσίας και ε, ιδιωτών, αύξηση του ΦΠΑ, ε, εισαγωγή νέων φορολογικών, οικολογικών συγγνώμη, φόρων και αύξηση των φορολογικών συντελεστών όπως στις φαρμακευτικές ε, υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, που είναι το 60% της προσπάθειας της οικονομικής εξεγείωσης, ε, εκεί μειώνονται τα επιδόματα ανεργίας, μειώνεται κατά 7% η κρατική προσφορά, μειώνουμε τις δαπάνες όλων των ε, Υπουργείων και φυσικά με βάση την τελευταία δημοσκόπηση είχαμε 230.000 ε, μείωση των δημοσίων υπαλλήλων και μείωση ε, κατά 23% των ε, φαρμακευτικών δαπανών μετά τη μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας. Σε ό,τι αφορά τις αυτόνομες κοινότητες, είχαμε σημαντικές, σημαντική πρόοδο στη διαφάνεια και τον έλεγχο των λογαριασμών τους, καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο των σχέσεων με τις αυτόνομες κοινότητες. Ε, φυσικά έχουμε την αρχή της δημοσιονομικής οροπίας ως συνταγματική αρχή, όπως προβλέπει ο Οργανικός Νόμος ε, ε, Δημοσιονομικής Σταθερότητας και ο νόμος αυτός θεσπίζει το πλαίσιο δημοσιονομικών σχέσεων μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των αυτόνομων περιφερειών. Σε ό,τι αφορά την διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, περάσαμε από την τρίμηνη στην μηνιαία ε, τακτικότητα. Έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με την εκτέλεση των λογαριασμών των αυτόνομων περιφερειών. Έχουμε επίγνωση ότι η οι εκτιμήσει που γίνονται διεθνώ για την Ισπανία στερούν σε σχέση με τι δικέ μα. Βέβαια, οι προβλέψει αυτέ ε, δεν είναι αδιάψευστε. Εμεί συνεχίζουμε τι ε, οικονομικέ μα μεταρρυθμίσει και τα προγράμματά μα για να υλοποιήσουμε τι δικέ μα προβλέψει που τι θεωρούμε ρεαλιστικέ. Αναφέρεται ότι το μέλλον του ευρώ θα κριθεί στην Ισπανία. Θα είναι καταλητικό ο ρόλο μα και όσο πιο γρήγορα υιοθετήσουμε τη, ε, διαχειριστούμε την κρίση του ευρώ, τόσο πιο γρήγορα η Ισπανία θα επανέλθει στον δρόμο τη ανάπτυξη και μάλιστα σε δύσκολο ευρωπαϊκό και διεθνέ πλαίσιο. Αλλά ήδη διαπιστώνουμε κάποιε θετικέ ενδείξει που δείχνουν ότι οι προσπάθειε διόρθωση των ανισορροπιών θα αποφέρουν και μεσοπρόθεσμα καρπού. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα που αφορούν ε, τη διόρθωση των ανισορροπιών. Καταρχήν σχέση με τον εξωτερικό τομέα είναι η περίτρανη απόδειξη των αλλαγών της οικονομίας μας. Γιατί διορθώνουμε το έλλειμμα μας ε, του ισοζυγίου πληρωμών, θα φτάσουμε στην ισορροπία φέτος. Ε, βέβαια είχαμε ένα έλλειμμα που ήταν η αιτία των προβλημάτων μας, 10% του ΑΕΠ το 2007. Σε σχέση με, πρόσβαση, με πρόσφατα στοιχεία, το πλεόνασμα ε, για το 2013 θα ε, ε, υλοποιηθεί. Θα καταλήξουμε σε πλεόνασμα εκεί που είχαμε έλλειμμα. Φαίνεται ότι όλες οι προσπάθειε μα αρχίζουν και αποφέρουν καρπού και στο ισοζύγιο πληρωμών. Έχουμε μάλιστα και διαθροτικέ αλλαγέ, διορθώνεται το ισοζύγιο το εξωτερικό με την αύξηση των εξαγωγών μα και το εμπορικό μα έλλειμμα που έχουμε απέναντι στην Ισπανία το μειώσαμε κατά 50% στο πρώτο εξάμεινο και οι εξαγωγέ μα αυξάνονται προ τη Γερμανία με ρυθμό άνω του 7%. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε ε, εμπορικό πλεόνασμα εκτό από την ενέργεια και τι υπηρεσίε χωρί να περιλαμβάνουμε και τον τουρισμό κάτι που αποτελεί παράδειγμα και απόδειξη του, βιομηχαν... του ισχυρού και ανταγωνιστικού βιομηχανικού μας ιστού. Σε ό,τι φορά τώρα τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης αγοράς εργασίας. Ανακτήσαμε μεγάλο τμήμα της απώλειας ανταγωνιστικότητας που διαπιστώσαμε μετά την εφαρμογή του ευρώ στην Ισπανία. Καταρχήν, ε, μετριάστηκε η αύξηση των ε, μισθών, κάτι που συνεχίζεται. Ε, σε ό,τι αφορά τα το κόστος μονάδας που είχε διαπιστωθεί από το 2009 μειώνεται και μάλιστα το 2012 θα έχουμε γύρω στο 100% το βασικό επιτόκιο, κάτι που δείχνει την ε, ανταγωνιστικότητα της ε, οικονομίας. Σε ό,τι αφορά την, την αριθμική αναπροσαρμογή των μισθών εξαφανίζεται και οι συμβάσεις με την αριθμική αναπροσαρμογή ήταν 28% το 2012 και μειώνεται. Σε ό,τι αφορά με τελευταία στοιχεία της δημοσκόπησης, ε, παρόλο που δεν είναι θετικά, έχουν δύο στοιχεία που κατά τη γνώμη μου ε, έχουν μεγάλη σημασία. Έχουμε σταθεροποίηση στην εξέλιξη των στοιχείων του ιδιωτικού τομέα και Βέβαια, η απώλεια θέσεων απασχόληση επηρεάζει κυρίω το δημόσιο τομέα. Εκεί γίνεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια εξυγίαση των οικονομικών. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν παράδειγμα ότι η εργασιακή μεταρρύθμιση δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο για τι εργασιακέ σχέσει. Το τρίτο στοιχείο, από την άποψη τη βελτίωση ε, των ανισορροπιών της ισπανικής οικονομίας είναι η ανάλυση των οικονομικών συνθήκων. Και παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στις κεφαλαγορές, σήμερα έχουμε, ανακτήσει, έχουμε καλύψει πάνω το 100% των ταμιακών μας αναγκών για το 2012 και μάλιστα το, κόστος, το μέσο κόστος των ισπανικών ομολόγων μένει στο ίδιο επίπεδο του 2011. Και μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την αγορά ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, δημιούργησε ένα νεωμένο και ζωηρό ενδιαφέρον των επενδυτών προς τα ισπανικά ομόλογα και αυξήθηκε το ποσοστό τους ε, φτάνοντας μέχρι το 35%. Η ισπανική οικονομία φαίνεται ότι ε, με ταχύς ρυθμούς ε, βελτιώνεται. Και η χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά μειώθηκε. Είναι κάτι που αντιστοιχεί στο 15% του ισπανικού ΑΕΠ. Όλα αυτά τα στοιχεία μα δείχνουν ότι η Ισπανική κυβέρνηση βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Έχουμε επίγνωση ότι οι προβλέψει, οι δικέ μα για την Ισπανία είναι πολύ πιο αισιόδοξε από τι εκτιμήσει των διεθνών οργανισμών. Παρ' όλα αυτά, κατά το πρώτο εξάμεινο, οι διεθνεί προβλέψει ευθυγραμμιζόταν σε μεγάλο βαθμό με τι δικέ μα. Κάναμε κάποιε προσαρμογέ τη φορά το ΑΕΠ του 2012, που αναμέναμε μείωση 1,7%, τώρα διαπιστώνουμε ότι είναι 1,5% και φαίνεται ότι το τελικό στοιχείο για το 2012 θα είναι ακόμη καλύτερο από τη μείωση του 1,5%. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κυβέρνηση είναι συνετή ως προς τις προβλέψεις της και κάνει μάλλον συντηρητικές προγνώσεις. Σε ό,τι αφορά το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο κινείται η ισπανική οικονομία, θα ήθελα να τονίσω ότι η ανάκαμψη της ισπανικής οικονομίας συνδέεται με την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και ιδιαίτερα με την κατάσταση στη ζώνη ευρώ μια ζώνη Ευρώπη που αντιμετωπίζει ύφεση και κρίση αξιοπιστίας εξαιτίας έλλειψης εμπιστοσύνης προς το ευρώ, κάτι που πειράζει όλα τα κράτη-μέλη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαβεβαίωσε ότι το σπρέτ της Ισπανίας είναι υψηλό, πολύ υψηλότερο από ό,τι θα έπρεπε και θα έπρεπε να είναι γύρω στο, ε, στις 200 ποσοστίες μονάδες, κάτι που επηρεάζει το κόστος χρηματοδότησης και του ιδιωτικού τομέα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι απαράδεκτο. Με βάση τις, τα, ε, τα στοιχεία της ΕΚΤ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ισπανίας πληρώνουν το διπλάσιο για ένα δάνειο από τις γερμανικές. Αν λύσουμε λοιπόν τα προβλήματα του ευρώ, θα επηρεάσουμε άμεσα και την ανάκαμψη τη ισπανική οικονομία. Τα κοινοτικά θεσμικά όργανα θα πρέπει να δώσουν αποδείξει για την βούλησή τους να καταλήξουν σε καλύτερη, μεγαλύτερη δημοσιονομική, τραπεζική και οικονομική ολοκλήρωση. Μόνο έτσι θα διέλθουμε από την κρίση. Ο μηχανισμό ε, εξαγορά ομολόγων στη δευτερογενή αγορά από την έκτη είναι θετικό όχι μόνο για την ε, δευτερογενή αγορά, γιατί δείχνουν αυτή τη σιδερένια βούληση ε, υποστήριξη του ευρώ, που είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Πιστεύουμε ακράδαντα στο ευρωπαϊκό όραμα και τηρούμε τις υποχρεώσεις μας ως μέλη της ε, Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι το ευρωπαϊκό όραμα και η ευρωπαϊκή οικοδόμηση είναι το καλύτερο δυνατό όραμα για την Ισπανία και για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Thank um, Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, το υπόλοιπο του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας, έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις προς τον Υπουργό. Θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε το πρότυπο του πεντάλεπτου. Μια ερώτηση και μια απάντηση, δηλαδή εντός πέντε λεπτών. Έχουμε πρώτα του ομιλητέ εξ ονόματο των ομάδων και μετά το, διαδικασία Catch the Eye. Και θα σα διαβάσω ποιου έχω σημειώσει, ώστε αν κάποιον ξεχάσαμε να αρχίσετε να ε, ζητάτε πάλι το λόγο. Ελκ. The S&D, it will be Sanchez Prozedo. For ALDE, it will be Ramon Tremosa. Do I detect some Spanish interest here? Uh... Κάπως ισπανικό ενδιαφέρον διαβλέπω εδώ. From Ava, uh, for the ECR we make a breakthrough with Dirk Effink. Um, then we come to... Και έπειτα στο Κατζιάι έχω. Betty Annie and Philippe Lamberts. Uh, others who want to be... Ποδηματά και If you wave, uh, more Spanish interest coming in. But anyway... Κι άλλο ισπανικό ενδιαφέρον βλέπω. Ο κύριος Άλμπα. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Ισπανό Υπουργό που ήρθε εδώ ως Ευρωβουλευτής και ιδιαίτερα Ισπανός. Αισθάνομαι ιδιαίτερη περηφανή για τις προσπάθειες που έκανε η Ισπανία και για την προσπάθεια που έκανε ο υπουργό να βρίσκεται σήμερα εδώ. Επίσης αναφερθήκατε στις άνευ προηγουμένου μεταρρυθμίσεις που ε, θέσπισε η Ισπανική κυβέρνηση και τονίσατε την ε, κεντρική μεταρρύθμιση που είναι η χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση, η δημοσιονομική μεταρρύθμιση. Μπορείτε να μας κάνετε μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής της μεταρρύθμισης και επίσης ε, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των τεστ αντοχής των τραπεζών θεωρώ ότι ένας από τους βασικούς στόχους αυτής της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της πατρίδας μας. Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να μας κάνετε και μια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ε, που έγιναν, ε, ε, των μεταρρυθμίσεων που έγιναν για την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Ευχαριστώ. Θα μπορούσα να μιλήσω αγγλικά, αλλά μια και η ερώτηση τέθηκε στα ισπανικά. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα και η απάντηση να δοθεί στα ισπανικά. Σε ό,τι αφορά την χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση, νομίζω ότι το σημείο φετηρίας, που δεν το τονίζουμε αρκετά μερικές φορές είναι το πρόβλημα αξιοπιστίας που υπήρχε απέναντι στην χρηματοπιστωτική θέση του Ισπανικού τραπεζικού συστήματο. Υπήρχαν αφιβολίε ε, για τα ισοζύγια, για του ισολογισμού των τραπεζών τη Ισπανία, Κάτι που είχε αρνητικό αποτέλεσμα, όχι για τις πιο ασθενείς τράπεζες ε, και οργανισμούς, αλλά ακόμη και για τους, ε, για τους φορείς που έχουν εξι, εξηγιαμένους υγιείς ισολογισμούς. Στόχος λοιπόν της κυβέρνησης ήταν από την αρχή να αποκαταστήσει τη διαφάνεια και την σαφήνεια των λογαριασμών στο ισπανικό τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα εν γέννη. Η Ισπανία λοιπόν εφάρμοσε καταρχήν, έκανε μια προσπάθεια άσκησης του, του stress, έκανε το stress test, το τεστ αντοχής, top-down, με βάση το, συστάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και έκανε ακόμη δύο τεστ ανοχής από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές. Και έγινε και κάτι άνευ προηγουμένου στην, στην Ισπανία. Είναι ένα αντίθετο stress test με αντίθετη μεθοδολογία bottom-up και έτσι αξιολογήσαμε σχεδόν το σύνολο του χαρτοφυλακίου, το 90% του ισπανικού τραπεζικού συστήματος. Τα σενάρια που προέβλεπαν αυτά τα τεστ αντοχής ήταν πολύ διαφορετικά. Αναμένονταν ΑΕΠ, μείωση ΑΕΠ πολύ μεγαλύτερο, ε, κάποιες ε, προσαρμογές ανεφροηγουμένου ε, και επίσης δινόταν ένας χρονικός ορίζοντας τριών ετών, ενώ τα, τεστ, τα stress test έχουν χρονικό ορίζοντα δύο ετών. Διαπιστώσαμε τελικά το 70% του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου είναι υγιές, κατά βάση, και παρά το αρνητικό σενάριο, οι ισπανικές τράπεζες έχουν ένα πλεόνασμα κεφαλαίου γύρω στο 70%, κάτι που ε, οδήγησε σε αποτελέσματα που δεν είχαμε στις γειτονικέ χώρες. Σίγουρα είμαστε η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία το τραπεζικό σύστημα και η τράπεζα ε, υπέστησαν τις μεγαλύτερες και τις πιο εξονυχιστικές αναλύσεις, αξιολογήσεις και εξετάσεις. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Τώρα, υπάρχει το θέμα της έγχυσης κεφαλαίου, δύο μέτρα χρειάζονται, η τροφοδότηση με κεφάλαιο. Περιμένουμε την έγκριση των σχεδίων αναδιάρθρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Επίτροπος Αλμούνια ανακοίνωσε ότι θα εγκρίνει τα σχέδια αναδιάρθρωση τέλη του μηνός, οπότε τα χρήματα θα εισρεύσουν αμέσως μετά. Και όπως είπα και προηγουμένως, ε, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διορθώσεις που θα γίνουν, τις προσαρμογές και μετά την αξιολόγηση του Όλιβερ Γουάιμαν, του ανεξάρτητου αξιολογητή, του stress θα είμαστε κάτω από 40 δις 35-40 ε, δις, δηλαδή 3,5% περίπου του Ισπανικού ΑΕΠ. Τώρα, όσο ό,τι αφορά αυτή την κακή τράπεζα που θα θεσπίσουμε, τα επισφαλή στοιχεία θα περάσουν στην κακή τράπεζα με σημαντική μείωση. Θα έχουμε μία διάρθρωση κεφαλαίου που πλειοψηφία θα έχει στο κεφάλαιο γύρω στο 55% ο ιδιωτικό τομέα. Και μάλιστα τις επόμενες μέρες θα δούμε πώς θα εισρεύσει ιδιωτικό κεφάλαιο στην διάθρωση χρηματοδότηση αυτή της κακής τράπεζας. Και φυσικά θα έχουμε σημαντική προσπάθεια χρηματοδότησης Πάντως ε, με την αποσαφήνιση αυτής τη διαδικασία. θα έχουμε ένα πολύ πιο υγιές τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ισπανία και με προϋποθέσεις για να χορηγούνται δάνεια. Ευχαριστώ Αντολίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας. Γνωρίζουμε ότι δεν έχετε εσείς όλες τις οικονομικές ευθύνες της κυβέρνησης. Εσείς είστε όμως πολύ έγκυρος εκπρόσωπος και της Ισπανικής κυβέρνησης και θα ήθελα να σας πω ότι οι Ισπανοί σοσιαλιστές στην κοινοβουλευτική ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών θέλουν να συμβάλλουν ώστε η Ισπανία και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επανέλθουν στον δρόμο της ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να ενισχύσουμε την ΟΝΕ προς όφελος όλων των συμπολιτών μας. Θα ολοκληρωθεί σε λίγο ένας χρόνος από τότε που αναλάβατε την κυβέρνηση. Τα στοιχεία είναι γνωστά, μας τα παραθέσατε κι εσείς. Ήδη παρατείνεται η οικονομική ύφεση, η ανεργία αυξάνεται, συρρυκνώνεται η πίστοση, τα δεν υπάρχει ρευστότητα, ούτε έχει επέλθει η αναμενόμενη εξυγίαση. Οι προοπτικές φαίνεται ότι επιδεινώνονται όσο περνάει ο καιρός. Γι' αυτό και υπάρχει και ένταση στην κοινωνία μας και αύξηση αυτής της έντασης. Διερωτώνται λοιπόν οι συμπολίτες μας. Οι θυσίες που έχουν κάνει έχουν κάποια αξία, αξίζουν τον κόπο. Γίνεται σωστή και δίκαιη κατανομή των υποχρεώσεων και των θυσιών ή μήπως επιβαρύνουν αυτές περισσότερα τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού. Νομίζω ότι με την παρουσία σας θα πρέπει να χύσετε φως στην κατάσταση αυτή. Θα ήθελα να κάνω δύο επίκαιρες ε, ερωτήσεις για την ε, Ισπανική κυβέρνηση και δύο που έχουν πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Είπατε ότι καλύψετε τις ανταμέικες σας ανάγκες για φέτος, δεδομένων των δαπανών. Ε, καλό θα ήταν όμως να δούμε αν θα αν θα προσαρμόσετε τις συντάξεις στο, στο κόστος ζωής, αν θα υπάρξει μια αριθμική αναπροσαρμογή των συντάξεων. Νομίζω ότι είστε ο μόνο άνθρωπος που μπορείτε να διαλύσετε αυτή την αφιβολία. Πιστεύετε ότι μπορεί η Ισπανία να γλιτώσει, να αποφύγει τη διάσωση και με υποπίες προποθέσει Ε, μπορείτε να μας βεβαιώσετε ότι δεν είστε διατεθειμένος να υπογράψετε μια λευκό επιταγή. Αυτό θα ήθελα να το διευκρινίσετε. Σε ό,τι αφορά την, ε, τον προσανατολισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής, έχω δύο ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι οι πολιτικές προσαρμογής και αυτά τα προγράμματα ε, τόσο ε, ε, δρακόντια βελτιώνουν ή επιδεινώνουν τα προβλήματα. Μήπως θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναθεωρηθούν αυτές οι πολιτικές της λιτότητας. Επίσης, τα προγράμματα χρηματοπιστωτικής ενίσχυσης, αν ε, κατευθύνονται προς τα κράτη-μέλη αντί για τις τράπεζες, τελικά θα επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος, κάτι που έρχεται σε αντίφαση με τις υπόλοιπες πολιτικές της Ένωσης. Ενώ ταυτόχρονα μετατρέπουν ε, το, εξωτερικό, το εξωτερικό ιδιωτικό χρέος σε εσωτερικό κρατικό χρέος. Θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα ε, άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών κατά τη γνώμη χωρίς να περνάνε αυτές από τις κεντρικές κυβερνήσεις. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις με τη σειρά που τις υποβάλλατε. Σε ό,τι αφορά το θέμα των συντάξεων. Γνωρίζετε κι εσείς θαυμάσια ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε μεταρρύθμιση μετατοπίζοντας από τα 65 στα 67 το συντάξιμο της ηλικία. Είναι μια μεταρρύθμιση που κατά τη γνώμη μου βαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση της παράτασης του συντάξιμου όριου ηλικίας. Κάτι που καθιστά πιο βιώσιμο το συνταξιοδοτικό σύστημα. Δεν έχω πρόβλημα να αναγνωρίσω κάτι που έγινε σωστά από την προηγούμενη κυβέρνηση. Τώρα, αυτό που ανήγγειλε η Ισπανική κυβέρνηση για τις ε, επόμενες ημέρες και εβδομάδες είναι να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το κέριο πρόβλημα της κοινωνικής μας ασφάλισης, που δεν είναι τόσο ε, το όριο ηλικίας ε, συντάξεων, αλλά η ευθυγράμμιση τη πραγματική ε, ηλικία συνταξιοδότηση με τη νομική. Γιατί η πραγματική είναι στα 63 αυτή τη στιγμή και όχι στα 65 που προβλέπει ο νόμο. Θέλουμε λοιπόν να πλησιάσουμε την πραγματική ηλικία συνταξιοδότηση με την νόμιμη ηλικία συνταξιοδότηση. Που με βάση τη μεταρρύθμιση που ενέκρινε η προηγούμενη κυβέρνηση, η σοσιαλιστική, θα παραταθεί για δύο ακόμη χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σε μια κοινωνία που το προσδόκιμο ζωή αυξάνεται, είναι σημαντικό να προσαρμόσουμε τι παραμέτρου και των συντάξεων στο προσδόκιμο τη ηλικία. Είναι παράγοντα βιωσιμότητα κάτι τέτοιο. Όπω ξέρετε, ε, προσαρμόσαμε τη μαριθμικά κατά 1% της συντάξει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το, την ερώτηση για την διάσωση την περίφημη. Εγώ όταν με ρωτάνε και στο Κοινοβούλιο αυτό λέω πάντα. Η αγορά εκ μέρους της ΕΚΤ ε, ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, αν αυτό θεωρείται διάσωση, τότε όπως όλοι ξέρετε μεταξύ του Αυγούστου και του τέλους του προηγούμενου έτους είχαμε μια τέτοια ε, διάσωση, γιατί η ΕΚΤ αγόρασε σημαντικό τμήμα κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Τώρα, θα ήθελα να πω καταρχήν ότι η ευρωπαϊκή κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτό το σύστημα αγορά ομολόγων στη δευτερογενή αγορά και μέρου ΕΚΤ είναι θετικό. Όχι τόσο για την αγορά καθ' αυτή, αλλά γιατί επιβεβαιώνει τη βούληση της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που είναι το πρωταρχικό οικονομικό θεσμικό όργανο της Ένωσης, στη δέσμευση της ΕΚΤ υπέρ του μέλλοντος του ευρώ. Έτσι, διαλύθηκαν οι αμφιβολίες ως προς ότι το ευρώ είναι μη αντιστρέψιμο και οι χώρες που επλήγησαν από τις αμφιβολίες αυτές ήδη με την ανακοίνωση της ΕΚΤ διαπίστωσαν μια βελτίωση στην κατάσταση. Το σύστημα OMT της αγοράς, δηλαδή ομολόγων στη δευτερογενή αγορά από την ΕΚΤ που υπέβαλε η ΕΚΤ, πιστεύουμε ότι αυτό το σύστημα και αυτή η πρόταση είναι πολύ χρήσιμη και πολύ θετική και σε σε μεγάλο βαθμό διασκεδάζει τις ανησυχίες και τις αμφιβολίες που, είχα, που πλανώντας την ατμόσφαιρα προς το μέλλον του ευρώ. Τώρα, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε καλύψει τις ταμιακές μας ανάγκες για φέτος και σε ό,τι αφορά τις ε, σχέσεις μας με τα θεσμικά όργανα τηρούμε τις ε, διατάξεις του υπερβολικού, της υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη Συμφωνία για το Υπερβολικό Χρέος και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Από αυτή την άποψη κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας και να εκπληρώσουμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις που απορρέουν από τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Κανένας δεν αφισβητεί σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο τις προσπάθειες εξηγήσεις και τις μεταρρυθμίσεις που υιοθέτησε η Ισπανική κυβέρνηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πιο ευρωπαϊκές, όπως είπατε, ερωτήσεις, μιλήσατε για την πιθανή τροποποίηση ε, της ε, προσέγγισης της οικονομικής πολιτικής ε, και τη χρήση της δημοσιονομικής πολιτικής. Καταρχήν, είναι σημαντικό ε, να, μειωθούν, να, μειωθεί το δημόσιο χρέος. Πέρυσι ήταν 9% στην Ισπανία, είναι υψηλό, θα πρέπει να μειωθεί. Φυσικά με λογικό, συνετό και δίκαιο τρόπο. Ο βασικός μας στόχος ήταν 4,4, μετά 5,3, μετά 5,8, έμεινε στο 6,3% τελικά ο στόχος μας για το δημόσιο χρέος. Βέβαια, δεν θα πρέπει να αμελούμε τη γενική ύφεση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό αυτές τις συνθήκες οι δημοσιονομικές μας προσπάθειες θα πρέπει να λάβουν υπόψη όχι μόνο τους ονομαστικούς όρους ε, του δημοσίου χρέους, αλλά και τους στόχους της διαρθρωτικής προσπάθειας. Σε ό,τι αφορά τώρα το, το θέμα του δημόσιου χρέους και, την, και η επίδραση ε, της ε, χρηματοδότησης των τραπεζών ε, στο δημόσιο χρέος ή στην αύξηση του δημόσιου χρέους. Η τροφοδότηση με κεφάλαιο, η έγχυση κεφαλαίου στην Ισπανία δεν θα ξεπεράσει το 3,5% του ΑΕΠ, του Ισπανικού ΑΕΠ. Δεν είναι τεράστιο το ποσό. Και πρόκειται για μια χρέωση, ένα δανεισμό που έγινε υπό ευνοϊκούς όρους. 12, ομόλογα με περίοδο χάριτος 10 χρόνια και με, με, με, με όρους ε, χρηματοδότης που είναι του μηχανισμού διάσωσης και όχι του μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και θα δούμε και φυσικά τι, τα, κεφάλαια θα υπάρχουν ε, ε, τη στιγμή της ε, έγχυσης του κεφαλαίου. Οπότε, για άλλες χώρες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κεφαλαϊκές ανάγκες ήταν πολύ υψηλότερε από τις ισπανικές σε σχέση με το ΑΕΠ, είναι σημαντικό να είναι άμεση η έγχυση κεφαλαίου. Στην περίπτωση όμως της Ισπανίας, αυτή η άμεση έγχυση κεφαλαίου θα είχε πολύ χαμηλότερη επίπτωση στο λόγο δημοσίου χρέους ΑΕΠ. Επαναλαμβάνω, είναι 3-3,5%. Οπότε είμαστε υπέρ και της Τραπεζικής Ένωσης, γιατί πέραν των δικών μας ισπανικών αναγκών, θεωρούμε ότι η Τραπεζική Ένωση είναι πολύ σημαντικό βήμα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη. Ευχαριστώ. Uh, πολύ. Λίγο παραπάνω κράτησε όμως αυτή η ερώτηση και απάντηση. Οπότε έχετε ήδη καλύψει δυο χρονοθυρίδες οι σοσιαλιστές. Ραμόν Τρεμόσα. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Έχω τρεις ερωτήσεις, πολύ σύντομες. Φάνηκατε πολύ αισιόδοξο σε σχέση με τις οικονομικές προβλέψεις ε, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι πολύ αρνητικές για την Ισπανία. Και από τότε που ήρθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009, διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι προβλέψει είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα από ό,τι η Ισπανική κυβέρνηση. Οπότε, τι θα γίνει αν είναι σωστέ οι προβλέψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2013-2014. Θα είναι σε θέση να επιστρέψει όλο το χρέο η Ισπανία ή μήπω θα πρέπει να ζητήσει αναδιάρθρωση του χρέου τη. Δεύτερον, ο ίδιο ο πρόεδρο Ντράγκη αναγνώρισε εδώ σε μια παρουσία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι και τα δύο LTROs που έγιναν πέρυσι δεν χρησιμεύσαν για την αύξηση της πίστοσης ε, ε, των τραπεζών στην Ισπανία. Τώρα όχι μόνο μειώνεται ο δανεισμός, αλλά έχουμε και μία διαρροή ε, των αποταμιεύσεων. Μειώνονται οι καταθέσεις. Έχουμε διαρροή και των καταθέσεων στην Ισπανία. Πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει ε, να αποφύγουμε ένα κλείσιμο των τραπεζών και θεωρείτε ότι η μπάνκια θα πρέπει να κλείσει. Σας ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος και άμεσος και θα ξεκινήσω από την τελευταία σας ερώτηση. Πιστεύω ότι η Μπάνκια είναι μια πολύ σημαντική τράπεζα στο ισπανικό τραπεζικό σύστημα και μετά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού που θα γίνουν προς την κακή τραπεζα και μετά την έχηση κεφαλαίου που θα γίνει, πιστεύουμε ότι και η Μπάνκια θα θα βρεθεί σε πολύ καλύτερη κατάσταση φερεγγιότητας και πιστεύω ότι με τη νέα διαχείριση που θα κάνει θα εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Σε ό,τι αφορά τα LTROs, αυτό που έκαναν ουσιαστικά τα LTROs ήταν να αντιμετωπίσουν το θέμα του funding, της ρευστότητας των τραπεζών. Στην περίπτωση της Ισπανίας, όπως είπα και προηγουμένως, φαίνεται σαφώς ότι το πρόβλημα δεν ήταν τόσο πρόβλημα ρευστότητα, αλλά πρόβλημα φερενκιότητας κάποιων τραπεζών. Και κυρίως ε, των τραπεζών που ελέγχονταν από το ΦΡΟΠ. Δηλαδή, από την Bank, η Μπάνκε, η Καταλούνια Κάισα, θα ξέρετε την περίπτωση, και την Νόβα Κάισα Γκαλήθια, καθώς και η Τράπεζα της Βαλένθια. Αυτές ήταν οι τέσσερις τράπεζες που είχαν περισσότερα προβλήματα και είναι περίπου το 90% της, ε, θα απορροφήσουν το 90% της έγχυσης κεφαλαίου που θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Αυτές οι τέσσερις τράπεζες. Και μπορεί με απόλυτους όρους η μπάνκια θα είναι αυτή που θα λάβει τα περισσότερα κονδύλια. Ε, σε σχετικούς όρους, αν κάνετε έναν απλό υπολογισμό, θα δείτε ότι ε, θα είναι και ε, άλλες ε, τράπεζες που θα λάβουν μεγάλες βοήθειες σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση του χρέους. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ε, σχέση αν για 0,8 αύξηση ε, πέσουμε έξω. Σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάσει κάτι τέτοιο την κατάσταση. Είναι πολύ αμεληταία η επιρροή και δεν πρόκειται να ζητήσουμε αναδιάρθρωση. Και θεωρούμε ότι οι δικές μας προβλέψεις, τα προγνωστικά της ε, Ισπανικής κυβέρνησης στηρίζονται σε συγκεκριμένες δράσεις και μεταρρυθμίσεις. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να αποφύγουμε με τις κυβερνητικές δράσεις ε, να υλοποιηθούν τα πιο αρνητικά σενάρια ή αρνητικές προβλέψεις. Και ναι, μεν θα υπάρξει μείωση ε, του ΑΕΠ, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι η μικρότερη δυνατή. Ξενόματος ε, των Πρασίνων Ευχαριστώ. Ακούγοντάς σας, ε, αποκόμισε την εντύπωση ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν ε, καλό μαθητή που θέλει να εντυπωσιάσει το δάσκαλό του ή μάλλον τη δασκάλα του, γιατί είστε ε, βασιλικότεροι του βασιλέως ή μερκελικότεροι της Μέρκελ. Θα ήθελα ως προς τις προτάσεις να κάνω το εξής σχόλιο. Μας παρουσιάσατε τα μέτρα που θεσπίσατε ή τα μέτρα που θα εγκρίνετε ως προς τις δαπάνες. Τι γίνεται όμως με τα έσοδα. Και εκεί υπάρχει θεμελιώδες πρόβλημα που αφορά τη φορολογική ευθύνη. Γιατί δεν προτείνουμε πιο άμεσα τρόπο το κλείσιμο το ΣΥΚΑΠ. Γιατί να μην εφαρμόσουμε πιο ενεργούς, ενεργές πολιτικές για τη φοροαποφυγή και, τη φορο... και την πάταξη φοροδιαφυγής. Έχουμε 2 εκατομμύρια φτωχούς στην Καταλωνία, αλλά έχουμε αύξηση κατά 83% των... της αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων. Ποιο πληρώνει αυτά τα μέτρα, ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Αναφερθήκατε και στις διαστάσεις ε, του, στεγαστικού κλάδου και των ενυπόθηκων δανείων. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο ε, δράμα των, ε, του στεγαστικού κλάδου είναι οι εξώσει οι κατασχέσει που εξωθούν ορισμένους ανθρώπους μερικές φορές σε αυτοκτονία από απελπισία. Δεν θα πρέπει να ανασταλούν ε, οι εκτελέσεις των κατασχέσεων και των εξώσεων. Επευλήθη σήμερα μια σχετική πρόταση στη Βουλή. Η ερώτηση είναι απλή. Τι πρόκειται να κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Δεγκίντος. Έχετε και Το πρόβλημα της Ισπανίας ε, από άποψη βιωσιμότητας των ε, εθνικών οικονομικών δεν είναι τόσο το βάρος των δημοσίων δαπανών που βρίσκεται κάτω από το κοινοτικό μεσόρο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι τα έσοδα είναι πολύ χαμηλότερα από το κοινοτικό μεσόρο. Και αυτό φυσικά σχετίζεται και με την ε, φοροδιαφυγή. Γι' αυτό και υιοθετήσαμε μια νέα ε, νομοθετική πρόταση για την πάταξη φοροδιαφυγής, ε, αλλά και υποβάλαμε ε, προτάσεις όχι μόνο για τη δημοσιονομική πολιτική, αλλά και για τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Φυσικά, με το σχέδιο πάταξης φοροδιαφυγής πιστεύουμε ότι θα αυξήσουμε τα φορολογικά μας έσοδα πολύ περισσότερο από ό,τι πέρυσι. Επίσης, γνωρίζετε κάλλιστα ότι πολλές φορές οι κυβερνήσεις απρόθυμα ε, έλαβε μη δημοφιλή, έργα, ε, ε, μη δημοφιλή μέτρα αύξησης φόρων. αύξησης φοροκινήτων, αύξηση του φορολογικού συντελεστή του ΦΠΑ, συμπερίληψη έξι οικολογικών περιβαλλοντικών φόρων. Έγιναν πολλές προσπάθειες λοιπόν και σε επίπεδο εσόδων και σε επίπεδο δαπανών. Φυσικά περισσότερες προσπάθειες κάναμε σε επίπεδο δαπανών που είναι το 60% και όχι σε επίπεδο εσόδων που είναι το 40% το, της δημοσιονομικής προσαρμογής και προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο δίκαιοι γίνεται. Αναφερθήκατε στο θέμα των κατασχέσεων και των εξώσεων στην Ισπανία που είναι ένα επίκαιρο θέμα. Θα σας ανέφερα μία προσωπική μου γνώμη με την άδειά σας. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ισπανία ένα εκατομμύριο κενά σπίτια. Ένα εκατομμύριο κενά διαμερίσματα ε, σπίτια. Οπότε η Ισπανική κυβέρνηση ε, με το Υπουργείο Οικονομικών και με τη συμφωνία του μεγαλύτερου κόμματο τη αντιπολίτευση, τη αντιπολίτευση, ε, θα φροντίσουμε να υιοθετήσουμε κάποια μέτρα και θέλουμε να υπάρχει συμφωνία κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Θέλουμε να λάβουμε μέτρα ώστε καμία καλόπιστη οικογένεια να μην μείνει χωρί ε, σπίτι εξαιτία τη κρίση, επειδή εξαιτία αδυναμία πληρωμή του ενυπόθηκου δανείου. Μάλιστα, ε, τα μέτρα που θα υιοθετηθούν σήμερα το βράδυ από την Τεχνική Επιτροπή αυτό το στόχο έχουν. Βέβαια θα πρέπει να αποφύγουμε κάποια ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Επαναλαμβάνω πάντως ότι η Ισπανική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομίας της Ισπανίας ε, θεωρούν ότι είναι απολύτω απαραίτητο κοινωνικά ε, να εξασφαλίσουμε ότι καμία ε, καλοπροαίρετη οικογένεια να μην μείνει χωρίς στέγη εξαιτία της οικονομικής κρίσης και θα λάβουμε μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ, εγώ δεν προετοίμασα την ερώτησή μου στα ισπανικά. Ε, γι' αυτό θα διακόψω και θα υποβάλω την ερώτησή μου στα αγγλικά δυστυχώς. Θα ήθελα να γνωρίζω, Υπουργέ, περισσότερα για, την σχέση μεταξύ της Βάνκη και κάποιων μεγάλων ισπανικών εταιριών στις οποίες έχει δώσει η Δάνεια, όπως η Μπέρια, η οποία πρόσφατα παρουσίασε πολύ απογοητευτικά στοιχεία. πρώτη μου ερώτηση, η Μπέρια θα μπορέσει να αποπληρώσει τα δανειά της. Δεύτερον, υπάρχουν άλλες εταιρείε που να βρίσκονται σε παρόμοια θέση ε, παράδειγμα, η η εφημερίδα Ελπαΐς παραμένει εν ζωή με απλήρωτα δάνεια και η ποδοσφαιρική ομάδα Μαντρίτ που αγοράζει ποδοσφαιριστές από ολόκληρο τον κόσμο με δάνεια δανεικά και αγύριστα τους αγοράζει. Δεν ξέρω πολλά πολλά εγώ για το ποδόσφαιρο, αλλά ξέρω πως το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο χωρίς τέτοιες αγορές θα ήταν μη ανταγωνιστικό. Και έπειτα, η μπάνκια, δανείζει αφαιρέγγιες εταιρείε, κάτι τέτοιο, δεν, θα, ε, ε, δεν μπορεί να λύσει όλους, να βοηθήσει όλους. Αν μια διάσωση λοιπόν της μπάνκια θα λύσει το πρόβλημα, ε, τότε περισσότερες ακόμα αιτήσει για διάσωση θα υποβληθούν, ε, για bailout. Κοιτάξτε, σας απαντήσω στα αγγλικά. Κοιτάξτε, έχετε εστιάσει την προσοχή σας στην μπάνκια και θα πρέπει να σας πω ότι η Μπάνκια Σύμφωνα με την ε, δοκιμή αντοχής που έκανε ανεξάρτητος αξιολογητής, χρειάζεται 24 δις ευρώ επιπλέον κεφάλαια. Να μπορέσει να ξεπεράσει ένα εξαιρετικά αρνητικό σενάριο. Χρειάζεται λοιπόν πολλά, και πολλά κεφάλαια. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω, πέρα από αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ως ε, ανέκδοτο, ότι είναι ότι η μπάνκη αφού μετέφερε τις τοξικές, ε, ε, τα τοξικά της στοιχεία στην κακή τράπεζα, στην bad bank και αφού θα λάβει τη βοήθεια που θα λάβει στις επόμενες δύο εβδομάδες, θα είναι ένα υγιές ίδρυμα πολύ σημαντικό για το τραπεζικό τοπίο της Ισπανίας. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι η διοικητική ομάδα, η διοικητική δίκηση μάλλον της Μπάνκια είναι πλήρω ανεξάρτητη και απόλυτα επαγγελματική. Η Μπάνκια πέρα από τα προβλήματα βραχυπρόθεσμης φερικαιότητας που μπορεί να αντιμετωπίζει Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό όνομα όσον αφορά την παρουσία, το δίκτυο ε, της, Μονάδε που έχει σε ολόκληρη την και ξεπερνά τι διάφορε αυτέ ε, ιστορίε και ανεκδοτά. Τώρα όσον αφορά την Ιμπέρια, η σχέση ανάμεσα στην Πάνκια και στην Ιμπέρια δεν είναι μια σχέση δανειστή με δανειζόμενο. Η Μπάνκια είναι σημαντικός μέτοχος της Ιμπέρια, νομίζω 30% αν δεν κάνω λάθος, και θα προσπαθήσει να μεγιστοποιήσει την αξία των μετοχών της στην Ιμπέρια με επαγγελματικό τρόπο. Um, e. Δεν είναι κανείς εδώ από την ΚΟΕ. E. Από το ΕΛΚ έχουμε τον κύριο Τεγκράντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν λέω καλώς ήρθατε στις Βρυξέλλες γιατί σχεδόν διαμένετε πια στις Βρυξέλλες όπως ε, και κάθε υπουργό που σέβεται τον εαυτό του ξέρει ότι στι Βρυξέλλε λαμβάνονται πολύ περισσότερες αποφάσεις και σημαντικές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την κοψότητά σα γιατί είπατε ότι η κατάσταση αυτή της κρίσης δεν ε, οφείλονται μόνο στην τελευταία κυβέρνηση, αλλά και στις προηγούμενες. Αλλά εσείς φυσικά καλείστε να την αντιμετωπίσετε. Σας ευχαριστώ και είχατε την κομψότητα να απαντήσετε ότι ε, γιατί η Μπάνκια δεν είναι μόνο θέμα Μαδρίτης, υπάρχει και η αντίστοιχη ε, τράπεζα της Βαρκελόνης. Προσπαθείτε, προσπαθεί η Ισπανία να τηρήσει τις προϋποθέσεις ε, που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί η κρίση τα θεσμικά όργανα βέβαια είναι τόσο άμεσα στις αντιδράσεις τους. Στο Συμβούλιο του Ιουνίου δημιουργήθηκαν μεγάλες υψηλές προσδοκίες, τονώθηκε η εμπιστοσύνη. Το επόμενο Συμβούλιο έκανε μία από τα ίδια και αυτή η κολυσιεργία, αυτή η βραδιπορία απελπίζει τους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί χρειάζονται κάποια μέτρα που θα είναι, είναι το αντίδοτο σε σχέση με τις θυσίες που έχει κάνει η Ισπανία και άλλες χώρες κατ' έτσι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Υπουργέ, κύριε Τεγκίντος, υπάρχει αναλογικότητα, υπάρχει αντιστοιχεία μεταξύ των θυσιών που κάνουν χώρε, όπω η Ισπανία, η δικιά μα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, με την ε, απελπιστική αργοπορία στη λήψη αποφάσεων εκ μέρου των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Υπάρχει τέτοια αντιστοιχεία. Ευχαριστώ κύριε Δεγκράντη. Θα έλεγα ότι και μπορεί να φαίνεται κάπω κατηγορηματική και ρητή αυτή η δήλωση, αλλά για την Ισπανία η οικονομική ανάκαμψη είναι πολύ δύσκολη και σχεδόν αδύνατη όσο δεν διασκεδαστούν οι αμφιβολίες ε, για το μέλλον του ευρώ. Γι' αυτό αυτό που θα κάνει η Ισπανία, πέραν το θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της ως προς την οικονομική της πολιτική, που φυσικά τη συντονίζει με, τη, με τους κοινωνικούς ε, εταίρους της και τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εξαρτηθούν πολλά από, το, από την Νομισματική Ένωση και την προσπάθεια διόρθωσης των προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο του ευρώ η Ισπανική κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι απαραίτητη και η Τραπεζική Ένωση και η δημοσιονομική ολοκλήρωση. Και επίση θα πρέπει να έχουμε ένα υγιές πλαίσιο ενιαίου νομίσματος και φυσικά δεν είναι μόνο η νομισματική πολιτική που είναι σημαντικές εδώ, αλλά και η δημοσιονομική πολιτική και άλλες πολιτικές που πειράζουν την ανταγωνιστικότητά μας. Και η θέση αυτή που είναι σαφώς υπέρ της ολοκλήρωσης και υπέρ της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και υπέρ του ενιαίου νομίσματος, υπέρ του ευρώ, μια τέτοια προσέγγιση θα μας ε, επιτρέψει να λύσουμε και τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα που έχει η Ισπανία. Σα είπα προηγουμένω ότι με βάση το Διεθνέ Νομισματικό Τομείο ε, χρησιμοποίησαμε και έναν ανεξάρτητο αξιολογητή. Με βάση το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, κανονικά το σπρέτ τη Ισπανίας θα έπρεπε να είναι 100 ποσοστιαίες μονάδε. Βέβαια η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική σήμερα όπω ξέρετε. Εξαιτία ακριβώ των αμφιβολιών που πλανώνται για το μέλλον του ευρώ. Θα είναι δι... διτή λοιπόν η προσπάθεια τη Ισπανίας. Θα κάνει ό,τι, ό,τι χρειάζεται και θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της στο εσωτερικό και θα προωθήσει ταυτόχρονα τις ε, θεσμικές μεταρρυθμίσει που χρειάζονται για να διασκεδαστούν οι ανησυχίε ω προς το μέλλον του ευρώ. Ευχαριστώ. Hey, um, I'm going to... Μάλιστα, θα προχωρήσουμε λοιπόν τώρα για... στον κύριο Λάμπερτς από του πράσινου και μετά θα επανέλθουμε στους Ελδημοκράτε. για να έχουν θέσει και αυτή τη ερωτήση. Ο Φιλίπ. Κύριε Υπουργέ, Καλησπέρα σας. Ε, μπορώ να σας μιλήσω στα γαλλικά. Κοιτάξτε, είχα την εντύπωση ε, ότι απευθύνεστε στη Bundestag ε, και μάλλον κακότυχο είστε γιατί ούτε Γερμανός δεν υπάρχει εδώ. σαν να θέλετε να δώσετε απολογισμό καλή διαγωγή. Εγώ θα σας δώσω αριθμητικά σε ερωτήσεις. Πρώτον, ποια είναι η, εκτίμησή σα για τις ε, δάνεια του, των Ισπανικών τραπεζών έχουμε ακούσει για 40 δις, για 60 δις, για 230 δις. Δεν ξέρω ποια είναι τα νούμερα της ανακεφαλοποίησης που θέλει να φτιάξει η Ισπανική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αλλά αν δούμε για 10, τα επόμενα 10 χρόνια, κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το σύνολο των απολειών που θα πρέπει να αναμένουμε ακόμα στον Ισπανικό τραπεζικό τομέα. Έπειτα, ε, υπάρχει όλη αυτή η αντίφαση ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Κομισιόν όσον αφορά το πολλαπλασιαστικό ε, παράγοντα των δημοσίων δαπανών στο ΑΕΠ. Για την Ισπανία, ποια είναι η δική σας εντύπωση για τον πολλαπλασιαστή. Έπειτα, ε, τελευταία ερώτηση. Πόσο καιρό θα κρατήσει ακόμα η Ισπανία χωρίς βία με έναν ποσοστό ανεργίας των νέων 51% και είπατε για τη στέγαση γιατί, ότι θα πρέπει να καθυστερήσουν ή να αποφευθούν οι ε, ξώσεις αφού υπάρχει ένα εκατομμύριο ε, κατοικίες που δεν, δεν είναι κατελημένες αυτή τη στιγμή. Άμα μείνουν άδεια αυτά τα σπίτια θα αρχίσουν να γκρεμίζουν. Δεν θα έπρεπε να αφήσετε να μπουν όλοι οι Ισπανοί που τα χρειάζονται σε αυτά τα αδιανά ε, σπίτια. Κοιτάξτε, τρεις ε, βασικές ερωτήσεις ε, σε σχέση με, θα απαντήσω στην τελευταία πρώτα, το 51% για τους νέους είναι πραγματικά παράδεκτο. Θα πρέπει να σας πω ως προς αυτό ότι η προηγούμενη νομοθεσία που είχαμε στην Ισπανία εστίαζε της την προσαρμογή των ισπανικών επιχειρήσεων, όποτε είχαμε ε, παραπάνω δραστηριότητα σε προσωρινά σε συμβάσεις, ε, δηλαδή τους, ε, τα outsiders της αγοράς εργασίας θα λέγαμε. Αυτό που θέλουμε τώρα μέσω της μεταρρύθμισης της αγοράς μας είναι ε, να εξαλείψουμε αυτή την αδικία, δηλαδή να αποφευθούν όλες ε, οι, προ, οι προσπάθειες προσαρμογής που κάνουν ε, οι εταιρείε, όταν δηλαδή έχουμε μία μείωση δραστηριότητας ή μείωση της ζήτησης, να επηρεάζονται αυτές οι συμβάσεις. Και γι' αυτό και έχουμε γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στους outsiders και τους insiders, δηλαδή τους συμμετέχοντες στην αγορά εργασίας Πολύ καλά, καλύτερο είναι κάποιε φορέ να προσπαθούμε να αποφύγουμε τις συγκρούσει και να έχουμε πολύ μεγαλύτερη ευελιξία ως όσον αφορά τις εταιρείε μας. Αυτό είναι ο βασικός στόχο στόχος της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας που εγκρίθηκε στην Ισπανία. Από την άποψη λοιπόν της Ισπανικής κυβέρνησης η νεανική ενεργεία θα είναι ο βασικός μας στόχος ε, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κοινωνική κατάσταση στη χώρα μας. Ε, πιστεύουμε ότι με 50% νέους άνεργους είναι αδύνατον να προχωρήσει μια χώρα και να προοδεύσει όσον αφορά την κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό λοιπόν θα εστιάσουμε την προσοχή μας και έχουμε γκρίνει μια νέα σύμβαση για τους νέους ε, την περασμένη μόλις εβδομάδα και όχι μόνο για να συνδυάσουμε μόνο την απασχόληση αλλά και να βασιστούμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο των νέων. Δηλαδή να προβλέψουμε την ε, κατάρτιση και την παιδεία των ανθρώπων με τη βαθμολογία. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό νέων στην Ισπανία που δεν είναι μόνο άνεργοι, είναι και εκτός της αγοράς εργασίας, ακόμα χειρότερα δηλαδή. Σε σχέση τώρα με τον πολλαπλασιαστή, είναι ένα θεωρητικό ζήτημα, το οποίο έχει ε, προκαλέσει, έχει μάλλον ε, τραβήξει την προσοχή και στα τελευταία συμπεράσματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είδαμε ότι ο πολλαπλασιαστής είναι τελικά ψηλότερος. Επηρεάζει περισσότερο από ό,τι είχαμε υπολογίσει πριν από τρεις-τέσσερις μήνες. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει κανείς υπόψη όχι μόνο την την, διαφθορωτική ε, προσπάθεια εξυγίασης στο οικονομικό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την, ε, τον κύκλο και να λάβουμε υπόψη όχι μόνο την ονομαστική μείωση του δημοσίου χρέους, αλλά και ε, από τη διαρθρωτική άποψη τη μείωση του χρέους και νομίζω πως η Κομισιόν τον λαμβάνει αυτό υπόψη. Και τέλος, η δοκιμή αντοχής που έγινε είναι δημοσιευμένη από την Τράπεζα της Ισπανίας και από το Υπουργείο Οικονομίας και μπορείτε να αναλύσετε τις ε, προτάσεις ε, και τις προεκβολές για απώλειες. Ε, είναι πολύ ε, ε, επικίνδυνο να προβλέψει κανείς σε προβλέψεις σε τέτοιες εποχές από τη στιγμή της κρίσης όμως αυτό που μπορώ να σας πω είναι και ότι παρά το γεγονός ότι στην Ισπανία λάβαμε πολύ αυστηρά μέτρα η προσπάθεια της στήριξης των ισπανικών τραπεζιζών ήταν τεράστια, ε, κοντά στο 12% του Ισπανικού ΑΕΠ, ώστε να κλείσει το χάσμα του χρέους που είχαν συσσωρεύσει οι τράπεζές μας. Για να δείτε δηλαδή ποια προσπάθεια έχουν καταβάλει έπειτα η κεφαλιακή ένες που θα δώσουμε θα είναι 3,5 του ΑΕΠ τελικά. Δεν είναι τόσο πολύ όσο σε άλλες χώρες ή όσο πιστεύουμε ή προβλέπαμε πριν από 6-7 μήνες. Νομίζω όμως ότι η βασική αξία όταν αναλύσει κανείς την κατάσταση, την κατάσταση του τραπεζικού τομέα της Ισπανίας είναι, να είναι ότι τελικά είδαμε πως η κατάσταση ήταν πολύ καλύτερη από την εικόνα που είχαμε αρχικά για την κατάσταση. Η κυρία Ποδηματά τώρα. Σας ευχαριστώ Σάρων, σας ευχαριστώ Υπουργέ για την πολύ λεπτομερή σας εισαγωγική ομιλία. Για να θέσω τα πράγματα λίγο διαφορετικά από τους προηγούμενους ομιλητές, θα ήθελα να σας ομολογήσω ότι όσο μιλούσατε, κατά το πρώτο τμήμα της εισαγωγικής σας ομιλίας, στράφηκα προς τον συνάδελφο Αντολίνα και του είπα ότι έχω την αίσθηση ότι ακούω τον Έλληνα Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Όχι ότι είναι συγκρίσιμη ασφαλώς η Ισπανία και η Ελλάδα, αλλά επειδή το μείγμα των πολιτικών, τα μέτρα τα οποία περιγράφεται σε ό,τι αφορά την μείωση των δαπανών, την αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όλα αυτά ε, αποτελούν τμήματα της συνταγή αν θέλετε. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθω στο ερώτημα του κυρίου Σάντσες Πρεσέντο. Ξέρω ότι καμία χώρα δεν μπορεί να τροποποιήσει αυτές τις πολιτικές ε, από μόνη της, αλλά δεν πιστεύετε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αλλάξουμε και να δώσουμε μια νέα ισορροπία σε αυτές τις πολιτικές, γιατί αναφέρετε και εσείς ο ίδιος την ύφεση η οποία επικρατεί σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαία, ξέρετε, αποτελεί απόρρια των περιοριστικών πολιτικών που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη. Και επιπλέον, Υπουργέ, και εσείς ε, αναγνωρίσατε το ποσοστό ανεργίας το οποίο είναι απαράδεκτο στην ε, Ισπανία. Το συνδέεται με τις ε, οικονομικές και κοινωνικές ανισορροπίες. Θεωρώ ότι ένα από τα βασικά αποτελέσματα των ανισορροπιών αυτών είναι ότι δεν υπάρχουν περιθώρια λιγμού στην τελική ανάλυση προκειμένου να υποστρέχθει η ισπανική οικονομία. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή και κατά δεύτερον Ποιοι, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί προκειμένου να βοηθήσουν την ανάκαμψη της οικονομίας στην Ισπανία. Απάντηση. Καταρχάς, δεν πρόκειται να κάνω οποιαδήποτε σύγκριση της ισπανικής οικονομίας με ε, οποιαδήποτε άλλη χώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό θα ήταν ε, προκατελημένο, επιτρέψτε μου να πω θα ήμουν ασφαλώς υπέρ της ισπανικής οικονομίας ε, προκατηλημένος. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Η ισπανική οικονομία είναι ανταγωνιστική, πραγματικά ανταγωνιστική. Αυτό προσπάθησα να το τονίσω και στην εισαγωγική μου ομιλία. Φέτος θα είμαστε πολύ κοντά σε μια ισοζυγισμένη εξωτερική θέση. Αλλά αυτό αποτέλεσε το βασικό πρόβλημα της Ισπανίας στο παρελθόν. Τρεις βασικές ανισορροπίες έχουμε στην Ισπανία. Καταρχάς, ο, δημόσιο, ο ιδιωτικός τομέας. Κατά δεύτερον, η φούσκα των ακινήτων. Και τρίτον, η απώλεια ανταγωνιστικότητας, η οποία συσσωρεύτηκε μέχρι το 2008. Και ο συνδυασμός των τριών αυτών παραγόντων, σε συνδυασμό με την νομοθεσία για την αγορά εργασία. προκάλεσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Άρα η προσέγγιση της ισπανική κυβέρνηση είναι μία απόπειρα να αντιμετωπιστούν και να διορθωθούν αυτές οι ανισορροπίες. Αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ε, τραπεζικό τομέα μέσω σαφήνειας και διαφάνειας, μέσω αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης, προκειμένου να δοθεί νέα όθηση ε, ρευστότητας στην πραγματική οικονομία στο μέλλον. Κατά δεύτερον, προσπαθούμε να ξεπεράσουμε μια νομοθεσία για την αγορά εργασίας που είχε πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην κατάσταση των εργατικών δυνάμεων και ιδιαίτερα των νέων στην Ισπανία, όπως είπα και προηγουμένως. Και τέλος, προσπαθούμε να πάρουμε μέτρα για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη. Να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, να μειώσουμε τα εμπόδια εισαγωγής, να δημιουργήσουμε ανταγωνιστικότητα, να τροποποιήσουμε δομές, προκειμένου να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της ε, ισπανικής ε, οικονομίας. Και θα πρέπει να σας πω ότι αφορά την ε, οικονομική πολιτική, ότι για να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι κάτι εντελώς απαραίτητο, πραγματικά απαραίτητο. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω ε, ενός σωστού δρόμου, αν θέλετε. Νομίζω ότι πλέον όλοι είναι πεπισμένοι, σχεδόν όλοι είναι πεπισμένοι, ότι η οικονομική λιτότητα δεν οδηγεί πουθενά. Η λιτότητα αποτελεί ένα βασικό μεσοπρόθεσμο παράγοντα, αλλά θα πρέπει να είμαστε απόλυτα πεπισμένοι, θεωρώ, ότι χρειάζεται και σωστές δημοσιονομικέ πολιτικές. Θα πρέπει να μειωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα. Και αυτό θα πρέπει να γίνει. Είναι ε, εντελώ απαραίτητο και αναπόφευκτο. Αλλά θα πρέπει να γίνει και με τον σωστό λογικό τρόπο, με ένα ρυθμό μάλιστα που δεν θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα και εμπόδια στις εμπορικές δραστηριότητες. Και νομίζω ότι όλοι στην Ευρώπη κινούνται με αυτή την πεποίθηση. Ευχαριστώ, η Πρόεδρος, ο Γιώργο Φιέλ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ, Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Εγώ θα μιλήσω πορτογαλικά. Για να μην ε, πιστέψει κανείς ότι η Βυρική Χερσόνησο έχει μόνο ένα κράτος, θα μιλησω σιγά σιγά ώστε να με καταλάβετε καλά. Εγώ, όπως φαντάζεστε, παρακολουθώ από πολύ κοντά την ισπανική πραγματικότητα και συγκρίνω με τη δικιά μας πραγματικότητα της δική μου χώρας και θεωρώ πως υπάρχουν πολλά πράγματα που προχωρούν παράλληλα. Καταρχήν, ε, θα πρέπει να δούμε αν αυτά τα μέτρα εξυγίανσης ε, δεν δημιουργούν τεράστιες δυσκολίες για την μελλοντική ανάπτυξη των οικονομιών μας. Πώς γίνεται και στις δύο χώρες η ανεργία να έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Συμφωνώ με ένα συμπέρασμα το οποίο πρόσφατα παρουσιάστηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι για κράτη δηλαδή που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν δυσκολία και γιατί για να μπορέσουν να ξαναβρούν την ανάπτυξη, να ξεπεράσουν τα απλά θέματα δηλαδή τα διαρθρωτικά ε, ότι τα επιτόκια για αυτές τις χώρες θα πρέπει να είναι χαμηλότερα και οι όροι οι οικονομικοί ευκολότεροι, καλύτεροι. η διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε σήμερα. Δεύτερο, εσείς το πιστεύετε αυτό, δεύτερη ερώτηση, ε, αυστηρά ευρωπαϊκή, που έχει να κάνει με την Δημοσιονομική Ένωση που ε, πάει να δημιουργηθεί. Εσείς συμφωνείτε να υπάρχει ένας επίτροπος που να μπορεί άμεσα να επηρεάζει του εθνικού προπολογισμού. Σας ευχαριστώ και φυσικά μπορείτε να μιλήσετε, να μου απαντήσετε στα ισπανικά γιατί καταλαβαίνω τη γλώσσα σας. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, το είπα και εγώ προηγουμένως. Με βάση τα σχόλια του Διεθνούς Ομισβατικού Ταμείου και άλλους υπολογισμούς που κάνουμε, θεωρούμε ότι το σπρέ της Ισπανίας και τα επιτόκια που καταβάλει η Ισπανία για τον δανεισμό της θα έπρεπε να είναι κανονικά γύρω στις 200 ποσοστίες μονάδες. Αυτό το αναγνώρισε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όταν ε, υπέβαλε την πρόταση για την εξαγορά ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά. Διαπίστωσε ότι υπήρξαν ε, ε, ταραχές ανομαλίες ε, στην αγορά εργασίας. Είναι μια πραγματικότητα, είναι υπέρον κατά επιτόκια δανεισμό που καταβάλουμε. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα, υπολογίσαμε ότι με μια μείωση κατά 100 ποσοστιαίες μονάδες ε, στην καμπύλη επιτοκίων στην Ισπανία, θα οδηγούσε σε αύξηση της ανάπτυξης στην Ισπανία γύρω στο 0,5% του ΑΕΠ. Είναι χαρακτηριστικό της ευαισθησίας που δείχνει και του, πόσο τρωτή είναι η πραγματική οικονομία απέναντι στις εξελίξεις των επιτοκίων. Και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να εξαλείψουμε τις αμφιβολίες ως προς το μέλλον του ευρώ. Αυτό θα επηρεάσει θετικά α, την ανάπτυξή μας. Και επίσης πέραν ε, των κινδύνων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αποτρέψουμε τους κινδύνους του ευρώ. Γι' αυτό και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του ευρώ για μας είναι πολύ σημαντική και έχει κέρια σημασία. Το δεύτερο ερώτημά σας αναφέρεται στην πρόταση για τον υπερεπίτροπο. Εμείς είμαστε υπέρ της ε, δημοσιονομικής ολοκλήρωσης ε, και της μερικής εκχώρησης κυριαρχίας για την, δημοσιονομ... για την επίτευξη αυτής της Δημοσιονομικής Ένωσης, αλλά εκτός από το, το ρόλο του υπερεπιτρόπου, ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι αυτό που λέμε accountability, η λογοδοσία. Η ανάληψη της ευθύνης και η λογοδοσία είναι πολύ σημαντικό γιατί όσο περισσότερες αρμοδιότητες έχει ε, κάποιος τόσο μεγαλύτερη ευθύνη έχει και τόσο, τόσο πιο επιτακτική είναι η ανάγκη για checks and balances, για ισορροπίες και ελέγχους. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την Πορτογαλία, με την Ελίζα Φερέιρα. Ευχαριστώ. Όπως και ο προηγούμενο ομιλητή θα μιλήσω πορτογαλικά. Αλλά μπορείτε να μου απαντήσετε στα ισπανικά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ που είστε σήμερα εδώ. Πρώτη μου ερώτηση. Ποιε ακριβώς είναι οι ημερομηνίε και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την αρχή της ανάπτυξης της ε, ισπανικής οικονομίας και με την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Κύριε Υπουργέ, συνειδητοποιείτε ότι όλες οι χώρες διαρθρώνουν την ανάπτυξή τους με μια προοπτική εξαγωγών. Αλλά εφόσον όλοι κάνουμε, ακολουθούμε την ίδια λογική, διερωτώμεθα, μα ποιος θα αγοράσει όλες αυτές τις εξαγωγές. Δεύτερο ερώτημα. Δεν μιλήσατε για επενδύσεις και πιστεύω πως η ανάπτυξη απαιτεί επενδύσεις. Εγώ πιστεύω πως για την Ισπανία είναι πολύ σημαντική η... σημαντικά τα διευθυντικά ταμεία. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε πάνω στις δημοσιονομικές προπτικές για το 2014 και μετά. Ποια είναι η θέση της Ισπανίας σε σχέση με την, το γενικό όγκο των ταμείων αυτών και δεύτερη ερώτηση. Η Ισπανία δέχεται αυτό που ονομάζεται macroeconomic conditionality, ε, μακροοικονομική όρη δηλαδή. Ε, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα κοινοτικά ταμεία αν παραβιαστούν ε, οι όροι του χρέους, ε, του ελλείμματος κτλ, μπορεί τα διευθυντικά ταμεία να ε, περικοπούν ως τιμωρία. Συμφωνεί η Ισπανία. Και ποια είναι η θέση της στο Σύμβουλο. Ευχαριστώ σε ό,τι αφορά του κινδύνου για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ισπανία. Θα έλεγα και το είπα και προηγουμένως ότι αυτή τη στιγμή η Ισπανία, όπως και άλλες χώρες της περιφέρειας που ίσως θεωρούνται πιο ευάλωτες στο ευρώ, χρειάζονται μια εξομάλυση των, όρων χρηματοδότηση οικονομίας. Αυτό χρειάζονται όλες οι χώρες. Εμείς φέτος καλύψαμε πλήρως, ε, όπως είπα, τις ταμιακές μας ανάγκες, αλλά δεν μπορεί μια μικρομεσαία επιχείρηση Ισπανίας να έχει κόστος δανεισμού πολύ ψηλότερο από ότι μια μικρομεσαία ε, επιχείρηση του κέντρου της Ευρώπης που δεν έχει τέτοια προβλήματα τροτότητας γιατί δημιουργεί ε, συγκριτικό μειονέκτημα μια τέτοια κατάσταση για τις ισπανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το επισήμανε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φαίνεται ότι είχαμε παρεθνικοποίηση των το, ροών κεφαλαίων εντός της ΩΝΕ και τελικά καταλήγουμε σε μια νομισματική πολιτική που δεν είναι ενία γιατί δεν ε, ε, λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο τα επιτόκια της ΕΚΤ σε μια χώρα του σκληρού πυρήνα της ΟΝΕ από ότι σε μια χώρα της περιφέρειας που είναι πιο ευάλωτη. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, για να έχουμε ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων απασχόληση θα πρέπει πρώτα να ε, καταργήσουμε τις τεράστιες διαφορές μεταξύ των σπρέτ και των επιτοκίων δανεισμού μεταξύ των χωρών. Γιατί αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στις υποδομές. Όπως ε, είπατε κι εσείς, η Ισπανία ήταν ε, καθαρός δικαιούχος ενίσχυσης ε, τα τελευταία χρόνια και χρησιμοποίησαμε νομίζω πολύ καλά αυτές τις, ε, αυτά τα κοινοτικά κονδύλια. Και δείτε τις υποδομές στην Ισπανία βλέπετε ότι πραγματικά είναι σημαντική μοχλή επανόδου στην, στο δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης και της ανάκαμψης. Έχουμε πολλές υποδομές λοιπόν, αλλά ο βασικός τομέας επενδύσεων ήταν ε, ο κατασκευαστικός και αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει γιατί τώρα αντιμετωπίζει κρίση. Πριν από πέντε χρόνια είχαμε 700.000 ε, κατασκευές. Φέτος είχαμε πολύ λιγότερες. Θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που θα είναι λογικό. Ούτε στο επίπεδο του παρελθόντος που ήταν υπέρογκο, αλλά όχι και στο πολύ χαμηλό ε, επίπεδο κατασκευών που έχουμε σήμερα. Τώρα, τι θα αναζητήσουμε στο μέλλον. Θα αναζητήσουμε επενδύσει πολύ πιο συνδεδεμένε με τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε επενδύσει στο δυναμικό του, στην ικανότητά του, επενδύσει στη γνώση, στην τεχνολογία. Νομίζω ότι αυτές οι επενδύσεις θα είναι οι πιο επωφελεί. Σε ό,τι αφορά τι εξαγωγέ ε, που είπατε. Ακούω πολλές φορές ότι το κέρδος ε, της ανταγωνιστικότητας ε, δεν είναι κάτι ουδέτερο. Όλοι μπορούν να κερδίσουν σε ανταγωνιστικότητα όταν αυξάνονται οι εξαγωγές. Γιατί οι εξαγωγές του ενός είναι οι εισαγωγές του άλλου, αλλά και οι εισαγωγές δημιουργούν θέσεις απασχόλησης ε, που επίσης ε, μπορούν να τροφοδοτήσουν την ε, οικονομία. Δεν έχουμε λοιπόν, με την, ανταγωνιστικότητα, στην ανταγωνιστικότητα δεν είναι ο ένας κερδίζει και ο άλλος χάνει ή αυτό που κερδίζει ο ένας πρέπει κάποιος να το χάνει. Μπορούν όλοι να κερδίσουν και οι δικές μας εξαγωγές δεν γίνονται εις βάρος άλλων χωρών, της ανταγωνιστικότητας άλλων χωρών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές, η Ισπανία ήδη περνάει από κατάσταση του καθαρού δικαιούχου σε, στην κατάσταση του καθαρού συνεισφέροντα και μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούμε και ε, σε ένα πλαίσιο που η κοινή γεωρική πολιτική θα διδραματίσει και στο μέλλον πολύ σημαντικό ρόλο. Θα είμαστε λοιπόν αυστηροί και λυτοί και στον εθνικό μας προϋπολογισμό, θα είμαστε αυστηροί και στον κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά δυστυχώς οι χώρες του Νότου υφίστανται πολύ πιο έντονα την κρίση και η συνοχή, η γεωρική πολιτική διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για και θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη στο μελλοντικό προσδιορισμό των δημοσιονομικών προοπτικών. Ευχαριστώ. Κανένα άλλο μέλο δεν έχει. Θέλετε κάτι να προσθέσετε, μήπω. Γιατί θέσατε ένα ερώτημα και με συγχωρείτε γιατί το ξέχασα και δεν το απάντησα σε ό,τι αφορά τα και να, σπίτια στην Ισπανία. Αυτό που έχω να πω είναι το εξή. Βλέπουμε ότι έχουν προσαρμοστεί οι τιμέ ε, των ακινήτων προς τα κάτω στην Ισπανία. Ελπίζω δε ότι η τάση αυτή θα επιταχυνθεί και έτσι θα γευρώσουμε το χάσμα μεταξύ των τιμών της αγοράς και των τιμών που υπήρχαν σε κάποιους τομείς των ακινήτων ως τώρα. Αλλά κοιτώντας την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων της περιουσίας στην Ισπανία, θα καταλάβετε ότι σε κάποιους τομείς υπάρχει ήδη ε, καθοδική τάση και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό για την αγορά. Αυτή η μείωση των τιμών θα βοηθήσει τον κόσμο να είναι σε θέση να αγοράζει σπίτια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να συμβεί και θα πρέπει παράλληλα να διατύφονται και πιο πολλά δάνεια για αγορά ακινήτων προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση, ιδιαίτερα στους νέους. Ναι, Φίλιπ, ε, λέει η Πρόεδρος, έχει θέσει, έχει ζητήσει το λόγο ένα άλλο μέλος. Γκερέρο ζήτησε το λόγο. Έχω πρόβλημα με τα μάτια μου σήμερα. Ευχαριστώ. Κύριε Δεγίντο, και εγώ θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την παρουσία σα εδώ σήμερα και για τι πληροφορίε που μα δώσατε. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ανεργία. Τα στοιχεία του Οκτωβρίου ήταν δυσάρεστα. Ε, η Ισπανική κυβέρνηση και εσείς ο ίδιος σήμερα μας είπατε ότι η καλή είδηση, ή μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, η όχι τόσο κακή είδηση, είναι ότι η ανεργία επικεντρώνεται κυρίως στο δημόσιο τομέα, αλλά αυτή η είδηση κατά τη γνώμη μου είναι ε, διπλώς κακή, γιατί είναι συνέπεια της πολιτικής λιτότητας που εφάρμοσε η διοίκηση ε, και δεύτερον, επικεντρώνεται στις δράσεις ε, της ε, δημόσιας διοίκησης που αφορά, αφορούν παροχή υπηρεσιών και αγαθών σε πολίτες, δηλαδή στην παιδεία, στην, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στη δημόσια υγεία. Εκεί έγιναν οι περικοπές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, που καταρχήν θα είναι συνενετική. Δεν θεωρείτε ότι χρειάζεται κοινωνικό διάλογο για να αποφευθεί αυτή η καταστροφή των θέσεων απασχόληση ε, ε, στη δημόσια διοίκηση, στο δημόσιο τομέα. Επίση, ε, παρά τι ικανότητέ σα, φαντάζομαι καταλάβατε Πλήρω την ε, ερώτηση του συναδέλφου που είναι από τη Γαλλική αλλά ήταν πολύ ακριβής. Δεδομένων των ε, στοιχείων του πληθωρισμού του Νοεμβρίου θα κάνετε τη αριθμική αναπροσαρμόγη των συντάξεων για να αντισταθμίσετε την ε, απώλεια εισοδήματο σχέση με την αύξηση του 1% που εγκρίνεται στι αρχές του έτους και τη... την αύξηση του πληθωρισμού που προκύπτει από τα στοιχεία του Νοεμβρίου. επαναλαμβάνω, έγινε τη αριθμική αναπροσαρμογή των συντάξεων. 1%. Περιμένουμε ακόμη τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Νοεμβρίου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει νομοθεσία που ισχύει για το θέμα αυτό. Εν μέρει απάντησα στην ερώτηση του κ. Πρεσέδο. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο η μέσο και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συντάξεων. Και κατά τη γνώμη μου εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε και είπα ότι η σταδιακή παράταση του ορίου συνταξιοδότηση είναι πολύ θετική. Αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή πολύ περισσότερο είναι να ε, αντιστοιχίσουμε την πραγματική, ε, το πραγμα, την πραγματική ηλικία συνταξιοδότηση με την νόμιμη ηλικία συνταξιοδότηση. Γιατί υπάρχει χάσμα αυτή τη στιγμή. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε μέσω και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστήματος. Κοιτάξτε, όπου και αν χάνονται θέσει απασχόληση, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, η είδηση είναι κακή. Βέβαια, με βάση τα στοιχεία των δύο τελευταίων ε, ε, εξαμήνων, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση της απώλειας θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ενώ στον δημόσιο τομέα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ε, απώλεια θέσεων απασχόλησης εξαιτία των προσπαθειών ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης. Σίγουρα θα πρέπει να εξορθολογήσουμε τη δημόσια δίκη στην Ισπανία και σε κεντρικό και σε επίπεδο περιφερειακής αυτονομίας. Αυτό είναι, αυτός είναι ο στόχος, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μειώσουμε και το ε, δημόσιο έλλειμμα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στην κατάσταση αυτή και δίνω πολύ συχνά το εξή παράδειγμα. Γνωρίζετε ότι στην Ισπανία το 2007 είχαμε 2% ε, πλεόνασμα και κάτω από 40% λόγω δημοσίου χρέους και ΕΠ. Το 2009 περάσαμε δημόσιο, από δημόσιο έλλειμμα 11% και αυξήθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες ο λόγος ε, δημοσίου χρέους ΑΕΠ. Ξέρετε πώς ε, ε, εξελίχθηκε η ανεργία στην Ισπανία από το 2007 στο 2009. Από το 8% το 2007 φτάσαμε στο πάνω από 20% το 2009. Τι θέλω να πω ότι οι πολιτικές ε, φορολογικές δημοσιονομικής εξεγείασης δεν δίνουν πάντα την λύση για την ανεργία. Πολλές φορές έχουμε προβλήματα χρηματοδότησης Γι' αυτό και λέω ότι καλό θα είναι να γίνει μία λογική μείωση του δημοσίου ελλείμματος στην Ισπανία. Αλλιώς τα προβλήματα χρηματοδότησης θα είναι πολύ πιο σοβαρά. Ευχαριστώ. Μία μικρή ερώτηση έχω να σας κάνω και εγώ και έτσι να κλείσουμε. Σε ό,τι αφορά τα κέρδη από τις αγορές ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εξ όσων κατάλαβα, τα κέρδη υποτίθεται ότι θα έπρεπε να επαναδιανεμηθούν από τις κεντρικές τράπεζες, τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και αυτό κατά εφαρμογή των συνήθων συνηθισμένων κανόνων. Αλλά υπήρξε και μία συμφωνία κυρίων γιατί κύριοι διευθύνουν τις κεντρικές τράπεζες ότι τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να επαναπατριστούν. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο 35 ε, δισεκατομμύρια περιμένει η κυβέρνηση. Αναρωτιέμαι τώρα λοιπόν κατά πόσον οι κεντρικές τράπεζες έχουν προβεί σε αυτή την επαναδιανομή στις χώρες που έχουν πληρώσει αρχικά τα επιτόκια. Αυτό θα συνέφερε την Ισπανία και κάποιους άλλους. Και αυτό αν δεν έχει συμβεί, ίσως θα έπρεπε να το υπενθυμίσουμε. Το εξετάζουμε, απάντηση. Εξετάζουμε την κατάσταση αυτή πολύ προσεκτικά, όπως φαντάζεστε, και θα γίνει σήμερα μία σχετική συζήτηση και για την Ελλάδα. Αλλά μου προκάλεσε κάποια έκπληξη, γιατί στην ε, περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου η Bank of England έχει τέτοιο κέρδος. Είμαι απόλυτα πεσμένος όμως ότι αν ε, εκλεχτείτε στο μέλλον στην διοίκηση της ε, Τράπεζας της Αγγλίας θα αξιοποιήσετε τα κέρδη αυτά και θα τα διοχετεύσετε στην οικονομία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κέρδη αυτά. Και αυτό το έχουμε υπόψη και σε ό,τι αφορά συγκεκριμένε χώρε σε συγκεκριμένε καταστάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρο. Ελπίζουμε τα χρήματα να διοχετευτούν εκεί που πρέπει, εντό τη Ευρωζώνη. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν προαποφασιστεί για το Ηνωμένο Βασίλειο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον χρόνο σας.

Συνάδελφοι, θα ήθελα να κάτσετε, αν θέλετε, γιατί έχουμε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα να συζητήσουμε με τον Επίτροπο. Είναι σημαντικά λοιπόν τα θέματα αυτά σε ό,τι αφορά τα θέματα τα στατιστικά. Δύο θέματα εξετάζουμε, τους εθνικούς λογαριασμούς και την ε, αναθεώρηση των ε, στατιστικών πλαισίων. Έχουμε και τον ε, εισηγητή μας. Θα δώσουμε τον λόγο στον Επίτροπο, θα ακούσουμε τις ερωτήσεις και μετά ο Επίτροπος θα μιλήσει για θέματα φορολόγησης. Αυτό ασφαλώς είναι όχι μόνο σημαντικό οικονομικό θέμα, αλλά και πολιτικό θέμα. Μεταξύ άλλων και λόγω της απόφασης των ε, 11 κρατών μελών να προχωρήσουν για τη δημιουργία ζώνης ε, ε, ελευθερίου εμπορίου. Έχουμε θέματα φόρο διαφυγής και ούτω καθεξής. Να μην καθυστερήσουμε λοιπόν άλλο, να δώσω το λόγο στον Επίτροπο και μετά θα ακούσουμε τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πολύ για την, αυτή, την καλή εισαγωγή. Αξιότιμα μέλη. Από ένα χρόνο ε, ανέλαβα την αρμοδιότητα για τα θέματα στατιστικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν καλή χρονική στιγμή να κοιτάξουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία, η ευρωπαϊκή στατιστική. Η Επιτροπή θέλει να δημιουργήσει ένα στατιστικό σύστημα ε, ανεξάρτητο, ισχυρό και αποτελεσματικό για την δημιουργία ανεξάρτητων στατιστικών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά Τη συνάντησή μας στις 22 Δεκεμβρίου πέρσι, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ε, διάφορες πρωτοβουλίες. Σημειώσαμε πρόοδο για να αυξήσουμε την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων. Να σας αναφέρω κάποια σημαντικά λοιπόν νομοθετικά μέτρα. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πρόταση για την διόρθωση του κανονισμού για τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία και είμαστε πεπισμένοι ότι η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων δεν μπορεί να διασφαλιστεί χωρίς να γίνουν θαραλέες αναδιαρθρώσεις και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την άποψη αυτή και αυτό κατέστησε σαφές σε, σε θέματα ε, ελέγχου ποιότητας τα οποία ε, εγκρίθηκαν στις 13 Μαρτίου. Και επίσης την πρόσφατη έκταση του κυρίου Τσικλούνα που συζητήθηκε από την Επιτροπή σας την προηγούμενη εβδομάδα. Και ιδιαίτερος να πω ότι είναι αυξημένη η υποχρέωση λογοδεσία των επικεφαλής ε, των στατιστικών υπηρεσιών και χρειάζεται πιο έντονη συνεργασία με υπηρεσίες ε, ελέγχου. Επίσης, ο κανονισμός ε, θα συζητηθεί με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία. Τα κράτη-μέλη ε, διστάζουν να αποδεχτούν αλλαγές στο εθνικό του σύστημα σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την επαγγελματική ανεξαρτησία των επικεφαλής και τον συντονιστικό ρόλο που έχουν για τα στατιστικά στοιχεία. Στις πιο πολλές χώρες αυτές οι δύο δεν παρουσιάζουν προβλήματα, αλλά θα πρέπει φυσικά τα ίδια πρότυπα να ισχύουν για, όλα τα, για όλες τις χώρες. Και αυτό θα το πετύχουμε μόνο μέσω νομοθεσίας, θέσπισης νομοθεσίας. Δεν θα πρέπει οι εθνικές ε, ιδιαιτερότητες να παρεποδίζουν αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα. Και επίσης θέλουμε δεσμεύσεις ε, αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων. Όλα αυτά θα πρέπει να προσυπογραφούν από όλες τις κυβερνήσει για να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των εθνικών στατιστικών τους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπήρξε μια πρόσφατη απόφαση της Eurostat που ενισχύει την επαγγελματική ανεξαρτησία της Eurostat καθώς και τον στονιστικό του ρόλο στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εφαρμόζουμε τα ίδια πρότυπα που αναμένουμε και από τα κράτη-μέλη. Εκ παραλίλου, η απόφαση αυτή απαντά στις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά την έκθεσή του που ε, δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο. Η νέα απόφαση για την Eurostat επίσης ενσωματώνει την δέσμευση για την αξιοπιστή των ε, στατιστικών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι θέτουμε ένα καλό παράδειγμα για τα κράτη-μέλη τα οποία ελπίζουμε να ακολουθήσουν με μια εθνική δέσμευση. Γεγονός που προς το παρόν δεν έχει συμβεί. Αλλά δεν έχουμε χρόνο και δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Θα πρέπει να υπάρξει ανεξαρτησία από πολιτική, από την πολιτική επιρροή. Και ξέρω ότι αυτό βρίσκει σύμφωνο και το Κοινοβούλιο αλλά και την Επιτροπή. Θα πρέπει να συμφωνήσουν και τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να διασφαλίσουν την ε, επαγγελματική ανεξαρτησία των στατιστικών υπηρεσιών, ακόμα και αν αυτό προαπαιτεί αλλαγές στη γενική οργάνωση και στο νομοθετικό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να μεταδίδει αυτό το μήνυμα προς το Συμβούλιο και ελπίζω αυτό να αποτυπωθεί και στα αυριανά συμπεράσματα του ΕΚΟΦΗΝ. Κατά τρίτον, ε, οι αποφάσεις για τα πρόστιμα σε ό,τι αφορά α, την α, ε, νοθεία των στατιστικών στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει νομική αρμοδιότητα για τη εξαγωγή ερευνών στα κράτη-μέλη όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια νοθεία στατιστικών στοιχείων. Η Eurostat επίσης έχει ενισχύσει τη συνεργασία της με τις άνωτοπες αρχές ε, ελέγχου στην Ευρώπη. Αυτό θα μεγιστοποιήσει την, ε, τα αποτελέσματα των ελέγχων ποιότητας. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει ένα νομικό πλαίσιο για τα στατιστικούς δείκτες σε ό,τι αφορά τις μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες. Οι στατιστικές διαδικασίες θα προταθούν μάλλον τις στατιστικές διαδικασίες ε, συντόμως. Αξιότιμοι βουλευτές, όλοι ξέρουμε ότι το τρέχον ε, πλαίσιο δεν ευνοεί μεταρρυθμίσεις που προαπαιτούν και προσπάθεια αλλά και πόρους. Αλλά τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για την καλύτερη ε, συνεργασία και τον καλύτερο συντονισμό. τα επόμενα έτη θα υποβάλει σχετικές προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να βελτιώσει την ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων και Προβλέπεται δεύτερος γύρος ε, peer reviews, αναθεώρησης από ε, σε ό,τι αφορά τον κώδικα ορθών πρακτικών στα πλαίσια του ESS. Ε. Έτσι, η τρέχουσα κατάσταση θα αξιολογηθεί και θα προταθούν δράσεις από όλους τους φορείς που συμμετέχουν. Πολύ προσοχή θα δοθεί στην ποιότητα των στοιχείων σε ό,τι αφορά τα ελλείμματα και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο της σε οποιαδήποτε κατάσταση θεωρήσει ότι είναι απαραίτητο. Επίσης θα προταθούν μακροπρόθεσμες λύσεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων για ένα σύστημα για τα δημοσιονομικά της Ευρώπης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά δεύτερον, θα συνεχίσω να προωθώ τα φιλόδοξα σχέδια τα οποία πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωση της του 2009 για την παραγωγή των ε, στατιστικών στοιχείων. Η εφαρμογή των καινοτόμων αυτών ε, αρχών περνάει στη φάση καταγραφής πιλωτικών μελετών και ε, διαβουλεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια θα προβεί σε νομοθετικές προτάσεις για ένα λειτουργικό πλαίσιο συλλογής, διανομής και αρχιοθέτησης των ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων και πιστεύω ότι μεσοπρόθεσμα, στη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση όλα αυτά θα καταστούν μέρος της, καθημερινής, της καθημερινότητάς μας. Το Ευρωπαϊκό Στατιστικό πρόγραμμα μέχρι το έτος του 2017 που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνάδει με το όραμα αυτό. Η εφαρμογή του θα αποτελέσει μια πρόκληση και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για τα κρατημέλη. μελη Ωστόσο, δεν θα σημειωθεί οποιαδήποτε πρόοδος χωρίς τέτοια προσπάθεια. Θέλουμε να ανταποκριθούμε στις ε, προκλήσεις αυτές με συνεκτικότητα και συγκεκριμένες δράσεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι ο ρόλος των στατιστικών στοιχείων έχει δραματικά αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δεν αποτελούν μόνο ε, βασικούς παράγοντες για την, τα πολιτικά μέτρα. Χρησιμοποιούνται και για benchmarking χωρών και benchmarking της οικονομικής τους απόδοσης. Όλο και πιο πολλά μέτρα οικονομικά βασίζονται σε στατιστικούς ε, δείκτες δεδομένης της δυναμικής των αγορών. Τα στατιστικά στοιχεία μπορούν να αλλάξουν την, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτό μια ολόκληρη χώρα. Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι αυξάνεται η πολιτική πίεση και η πίεση από το κοινό για τα στατιστικά στοιχεία. Αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των μελλοντικών ε, μεταρρυθμίσεων σε ό,τι αφορά την, το συντονισμό της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής ε, της Ένωσης θα αποτελέσει παράγοντα σημαντικό. Θα πρέπει να τεσφαλιστούν λοιπόν τα μέσα αυτά προκειμένου να είναι πάντα αξιόπιστα και ανεξάρτητα τα στατιστικά στοιχεία. Ενδεχομένως να καταστεί αναγκαία η εκ νέου μεταρρύθμιση του πλαισίου για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων σε ό,τι αφορά τα πλαίσια, το πλαίσιο μεγάλων θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε απαραίτητε ε, προτάσεις και σε όλες τις μελλοντικέ δράσεις μας υπολογίζουμε στην υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και έχω ένα κατάλογο των ομιλητών που έχουν ζητήσει το λόγο. κούλα. Mr. Is there anyone else who'd like to speak? Κανείς άλλος ζητά το λόγο. Okay. So, Mr. Slikuta, you'd like to start. Thank you, Commissioner, for touching on these. Uh, Σας ευχαριστώ, Επίτροπε, που αναφερθήκατε σε αυτά τα τόσο σημαντικά και λεπτά ζητήματα που μας απασχολούν εδώ στο Κοινοβούλιο. Καταρχήν, σημειώνουμε μια φράση που είπατε την οποία θεωρώ πολύ σημαντική. Ότι τα κράτη-μέλη φαίνεται να είναι πολύ απρόθυμα να δεχτούν αλλαγές στα ισχύοντα πλαίσια. Ε, αυτό τα λέει όλα. Συμφωνούμε όλοι λοιπόν ότι χρειαζόμαστε αξιόπιστε στατιστικέ και ότι, ότι, ότι όλο ένα και περισσότερο τι χρειαζόμαστε εφόσον ε, οι θύνοντε για την πολιτική και θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσει σωστέ. Σημειώνουμε τις πρόοδε που έχουν, ε, που έχουν ε, επιτευχθεί μέσα στον κώδικα διοντολογίας της στατιστικής από το 2005 και την ανάπτυξη του νομικού πλαισίου που διέπει την εκπόνηση και την διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών. Ωστόσο, μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις, η Ευρώπη αντιμετώπισε ένα πρόβλημα. Όχι μόνο μια χώρα. Εκτέθηκε. Παρά τις ρήτρες, τις στατιστικές εκπονήθηκαν με παραπλανητικό τρόπο. Είμαστε τώρα σε μια φάση όπου συζητάμε την έκθεση για να βελτιώσουμε την ποιότητα των στατιστικών και πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στο τομέα αυτό, διότι δεν είναι ότι επειδή έγινε μια φορά δεν θέλουμε να ξανασυμβεί μόνο, αλλά και ότι Το νέο εξαπλό και στη συνέχεια διπλό πακέτο δίνουν τώρα στην Κομισιόν την δυνατότητα να ενεργήσει από τη στιγμή που οι χώρες δεν ανταποκρίνονται στους στόχους, τους οικονομικούς και τους δημοσιονομικούς. Με τη βάση κάποιων στατιστικών και δικτών, λοιπόν, οι χώρες θα τιμωρούνται και θα τους επιβάλλονται ε, πρόστιμα τεράστιων ποσών με τη βάση αυτών των στατιστικών. Άρα λοιπόν προκύπτει αυτό το θέμα. Ποιος φτιάχνει αυτές τις στατιστικές. Ποιος είναι ο αδύναμος κρίκος. Δεν έχει νόημα να είναι πολύ ισχυρή στη Eurostat και ίσως ε, και οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Από τη στιγμή που τα ίδια τα στοιχεία δεν είναι τόσο ε, βέβαια, τόσο σίγουρα. Παρά λοιπόν να μιλάμε για την ανεξαρτησία της Eurostat και των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών, να φροντίσουμε ώστε να είναι πραγματικά ανεξάρτητες και στις ε, επόμενες μας ε, συζητήσεις που θα, που θα γίνουν ε, και τις τροπολογίες που θα κάνουμε την τέλος αυτής της εβδομάδας την επόμενη εβδομάδα το αργότερο έχουμε υπόψη μας να έχουμε υπόψη μας μάλλον ότι το, το σύστημα θα το οθήσουμε μέχρι όσο πάει εκτός και αν χρειάζεται πια αλλαγή της συνθήκης. έτσι ώστε να μην ενδιαφέρει πια καθόλου από το ευρωπαϊκό σύστημα της κεντρικής τράπεζας όπου είναι σε διαρκή επαφή με τις κυβερνήσεις και την Κομισιόν. μέσα στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι υπόλογοι στα κοινοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό. Όλοι ξέρουμε βέβαια ότι οι κυβερνήσει θα αντισταθούν σε αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να μας εμποδίσει από το να πιέσουμε ώστε να δημιουργηθεί αυτό το σύστημα που πιστεύουμε ότι θα δώσει την απαραίτητη εξαρτησία. Δεν θα πια καμιά παρέμβαση από τις κυβερνήσεις. Σε εθνικό επίπεδο οι κυβερνήσεις λοιπόν θα είναι υπόλογες στα κοινοβούλια όπως είναι και οι ε, ορκωτοί λογιστές στις ε, χώρες. Εφόσον ορίζονται από τον Υπουργό οι διευθυντές της ε, Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και δεν μπορούν να, και μπορούν να απολυθούν χωρίς να αιτιολογηθεί η απόλυση, τότε τον, με τον ίδιο τρόπο οι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν να, για να ελέγξουν ή να επηρεάσουν τις εργασίες. Θέλουμε λοιπόν και εμείς αυτό να το αλλάξουμε και να έχουμε μια ανισορροπία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα θέλαμε λοιπόν να ο επικεφαλής ε, να είναι σε τη θέση του για, δυο, για, για 7 χρόνια, για συγκεκριμένο πάση περιπτώσει χρονικό όριο. Ότι θα πρέπει να εγκρίνεται και από το Κοινοβούλιο, να δίνει το Κοινοβούλιο γνωμοδότηση για τους υποψηφίους. Και φυσικά ε, τελευταίο λόγο θα τον έχει η Κομισιόν, αλλά τουλάχιστον το Κοινοβούλιο να μπορεί να δίνει μια γνωμοδότηση. Έχουμε λοιπόν προτάσεις ε, που τις υποβάλλουμε μέσω της έκθεσης. και έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα ενισχύσει την ανεξαρτησία των στατιστικών υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Τώρα, το σύστημα που θα βασίζεται στην σόρευση δεν ξέρω αν μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ορθή διακυβέρνηση, για συγκεκριμένους δείκτες, για χρονικές σειρές που θα πρέπει να συλλέγονται σε διεθνές ε, πλαίσιο, ή πάση ευρωπαϊκό πλαίσιο και με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές, ε, ώστε να έχουμε συγκεκριμένο λογιστικό σύστημα, ε, έτσι ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Έχω έξι ερωτήσεις στον καταλόγο. Θα πάρω τις ομάδε, αλλά δεν θα σα δώσω όλες, γιατί ξέρω πως είναι δύσκολο να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση και κάποιε φορέ φορές ξεχνάμε. Εμεί θέλουμε όλοι να πάρουν ε, απαντήσεις. Ο κύριος Λάμπερτ. Καταρχήν να σας καλωσορίσουμε Επίτροπε, ως ήθεστε δεν είστε υπεύθυνο μόνο για τα, το τι αλλά και για τα S, τις στατιστικές που πολλοί εδώ θεωρούν κακιά λέξη. Επίση, πιστεύω πω οι περισσότερε ερωτήσει προέρχονται από την αριστερή πτέρυγα τη αιθούση και η δεξιά πτέρυγα δεν κροσοπείται και τόσο πολύ. Ε, ναι, το ξέρω, αλλά είναι λίγοι από την δεξιά μεριά. Ίσως λοιπόν θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τις στατιστικές που αντιτίθεται στις ιδεολογίες ε, της ε, δεξιάς. Γι' αυτό δεν λείπει η δεξιά. Για το στατιστικές, τις στατιστικές και το εξαπλό πακέτο έχω μόνο ένα πράγμα να πω. Ξέρετε ότι συνεχίζεται η ο αγώνας κατά τον, του, του συγκεκριμένου παθητικού, πρόβλεψης παθητικού. Έχουν ε, οι χώρες ε, όπως η Γερμανία με νύχια και με δόντια αγωνίζονται λοιπόν για κατά του, του παθητικού, της πρόβλεψης μάλλον παθητικού εγώ θέλω όμως να έχουμε αξιόπιστες στατιστικές επιτακτικής βάσης για όλα αυτού του είδους ε, τις ε, δεχόμενες υποχρεώσεις, τις προβλέψεις υποχρεώσεων ή εγγύσεων. Ε, θα... Το λέω αυτό γιατί κάποιες φορές η Κομισιόν όταν έρχεται σε αντίφαση με τη Γερμανία πάει σιγά σιγά, προσπαθεί να μην προσβάλλει κανέναν ε, αυτούς που είπε το αφεντικό σας ότι μας πληρώνουν. τους να μην τους ε, προσβάλλει, γιατί αυτοί μας πληρώνουν. Το αφεντικό σας το είπε, Επίτροπε. Κάτι ακόμα το οποίο είναι ε, πολύ σημαντικό όσον αφορά τις επιθυμίες των πρασίνων, αυτό το υπόθεση του να ξεπερνάμε το ΑΕΠ, να ξεπεράσουμε το ΑΕΠ ως μοναδικό γνώμονα, το μόνο δηλαδή μέτρο Ξέρω πως αυτό το συμφωνείτε κι εσείς. Τι να περιμένουμε, να περιμένουμε κάποια ανακοίνωση από πλευρά σας για το επόμενο χρόνο. Δεν το ζητάω για το 2012, γιατί δεν έχουμε πολύ καιρό. Τι να περιμένουμε, συνήθως λέμε ότι ό,τι δεν παίρνει κανείς και με, άρα ό,τι μετράει έχει ως στοιχείο. Το μόνο που μετράμε εδώ είναι η ανάπτυξη του ΑΕΠ εμείς. Αλλά ούτε αυτό δεν έχουμε. Μήπως θα έπρεπε να αρχίσουμε να μετράμε κάτι άλλο ώστε να έχουμε μια κάποια ικανοποίηση ότι κάποια στοιχεία θα τα πάρουμε. Γιατί άμα ελπίζουμε για ανάπτυξη του ΑΕΠ, <laughs> μάλλον θα είμαστε απογοητευμένοι τις επόμενες δεκαετίες. Ευχαριστώ. Κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Θέλω να κάνω ορισμένα σχόλια σε αυτά που υπόθηκε, υπόθηκαν και θέλω να κάνω μια ερώτηση αξιοποιώντας αν είναι δυνατόν δώστε μου την άδεια την ιδιότητά σας ως υπευθύνου για τα θέματα φορολογίας. Αν είναι εκτός ύλης δεν θα την κάνω την ερώτηση, θα μου πείτε. Για τα θέματα της στατιστικής. Κύριε Επιτροπέ, η συζήτηση ενδιαφέρονται αυτά που μας είπατε όπως και ο εισηγητής μας αλλά δεν ήταν παρόμοιες, παρόμοιες οι τοποθετήσεις περίπου σαν αυτές που κάναμε πέρσι. Η ίδια συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι γίναν κάποια βήματα. Οι δικέ μου παρατηρήσει λοιπόν για να ε, σας αποκαλύψω ας πούμε την οπτική είναι πρώτον ότι το θέμα αυτό δεν είναι καθόλου τεχνοκρατικό. Καθόλου τεχνικό θέμα, καθόλου μαθηματικό. Οι εγκύκλειες σπουδέ μου με επιτρέπουν να τα παρακολουθώ αυτά με ευχέρεια, αλλά η παρατήρησή μου είναι ότι είναι άκρος πολιτικό ζήτημα. Σε τι συνίσταται η πολιτική πλευρά όλης αυτή της υπόθεσης, βεβαίως να βελτιωθούν οι τεχνικές κτλ. Αλλά το πρώτο είναι, το είπε και ο συνάδελφος, να το πω εγώ ίσως με πιο σαφέστερο τρόπο, ό,τι θες να καταγράψεις, ό,τι ζητάς, αυτές, αυτές τις απαντήσεις θα πάρεις. Και η επιλογή των μεγεθών και των στατιστικών που ζητάς να καταγράψεις, να παρακολουθείς την αλλαγή, είναι πολιτική επιλογή. Γιατί δεν καταγράφονται άλλα πράγματα που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είναι η μεγάλη συζήτηση πώς καταγράφεται και τι περιλαμβάνεται στην, ε, στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Δεύτερη πολιτική πλευρά είναι, το είπε και ο κύριος Συγκλούνα, ότι στο επίπεδο της, το εθνικό, αλλά επιτρέψτε μου να πω και στο ευρωπαϊκό, η λεγόμενη ανεξαρτησία των στατιστικών υπηρεσιών είναι προσχηματική. Ο υπεύθυνο τη στατιστική υπηρεσία σε εθνικό επίπεδο διορίζεται από έναν υπουργό, από μια πολιτική εξουσία και προφανώς οι επιλογές έχουν κάποια κριτήρια. Για δε το ευρωπαϊκό, διασκεδάστε μου αν μπορείτε την εντύπωση ή την ερώτηση που σας είχα κάνει και πέρσι και μου είχατε δώσει μια απάντηση αλλά δεν με ικανοποιεί από το γεγονός ότι αν η Eurostat που προείσταται των υπηρεσιών στατιστικής όπως στο παρελθόν διαπιστωθεί ότι ανέχθηκε αλλοιωμένα στοιχεία ποιος έχει την ευθύνη. Ποια θα είναι η πολιτική ευθύνη του αρμοδίου επιτρόπου, γιατί δεν έχω κάτι προσωπικά με εσάς, αυτού που θεσμοθετημένα εποπτεύει της Eurostat. Υπάρχει πολιτική ευθύνη. Πού θα αναζητήσουμε τη ζημιά. Διότι αν ε, υπάρχουν αλλοιωμένα στοιχεία όπως ξέρετε και ξέρω πάρα πολύ καλά, από αυτά τα στοιχεία μπορούν να προκύψουν διαφορετικές πολιτικές και διαφορετικές δημοσιονομικές πολιτικές, πειθαρχίε, κυρώσει και ούτω καθεξής. Επομένως, το πολιτικό ερώτημα παραμένει ως έστω και αν θέλουμε να λέμε συνεχώς για την ανεξαρτησία των στατιστικών αρχών. Και η ερώτηση για τα θέματα φορολογίας, αν ε, θα θέλατε να μου απαντήσετε, επειδή είναι ένα επίκαιρο θέμα, διάβασα ότι στην Daily Telegraph ότι υπάρχει μια λίστα της HSBC. Next. All Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για να μην μπλέξουμε πάρα πολλά, γιατί θα μα κάνει δύο διαφορετικέ παρουσιάσει ο Επιτροπό. Αν θέλετε, Επίτροπε, να μα απαντήσετε σε αυτέ τι ερωτήσει και έχουμε και άλλε δύο ερωτήσει να ακούσουμε. Σα ευχαριστώ. Κύριε Σεκλούνα, νομίζω. Μας παρουσιάσετε νομίζω τα τελευταία οκτώ έτη στην έκθεση και συμφωνούμε σε ό,τι αφορά το μέλλον του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ασφαλώς. Μιλώντας για ευρύτερα, μεγαλύτερα θέματα, θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα να συζητηθούν στο πλαίσιο μελλοντικών μεταρρυθμίσεων των συνθήκων. Το ανέφερα αυτό και εισαγωγικά. Αυτό θα αποτελούσε ασφαλώς μία βασική αλλαγή. Αλλά στην παρούσα φάση νομίζω ότι σημαντικό είναι να γίνουν οι βελτιώσεις της νομοθεσίας που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδέες της έκθεσής σας. Προκειμένου να εγκριθεί ο κανονισμός. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο για το πλαίσιο της ανεξαρτησίας των Ευρωπαϊκών Στατιστικών Υπηρεσιών. Είναι σημαντικό λοιπόν να εγκριθεί το συντομότερο δυνατόν ο κανονισμός. Σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που έθεσε ο φίλος κύριος Λάμπερτς για τα contingent liabilities, τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Το θέμα αυτό στο πλαίσιο των ε, τρέχουσων συζητήσεων για το Ευρωπαϊκό Σύστημα για το 2010. Νομίζω ότι καταλήξαμε σε ένα καλό συμβιβασμό και τελικά εγκρίθηκε η συμπερίληψη των ε, συντάξεων στο σύστημα. Φυσικά, μιλώντας γενικότερα, όσο πιο πολύ είναι η διαφάνεια για οποιοδήποτε, για οποιασδήποτε υποχρεώσεις, είτε είναι ενδεχόμενε είτε όχι, τόσο το καλύτερο για την αξιολόγηση της κατάστασης. Να σας ρωτήσω, κύριε Λάμπερτς, ξέρω ότι το επίπεδο οριμότητας που έχουμε για, την, ε, για τις ε, συντάξεις είναι πιο υψηλό από τα άλλα επίπεδα για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και υπάρχουν ίδιες υποχρεώσεις για αναφορά αλλά μπορούμε να υπολογίζουμε σε εσά για να φέρετε στο ίδιο επίπεδο και τις άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Φυσικά, βρισκόμαστε σε φάση διαρκούς βελτίωσης της μεθοδολογίας που ακολουθούμε στους τομείς αυτούς. Και φυσικά θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Eurostat σε ό,τι αφορά την ε, ανάπτυξη της μεθοδολογίας αλλά εξ όσων καταλαβαίνω ήδη εργάζονται και αναζητούν βελτιώσεις ε, της μεθοδολογίας και σε άλλους τομείς, όχι μόνο σε αποχρεώσεις για τις ε, συντάξεις. Για το θέμα τώρα του πέραν του ΑΕΠ. Να πω ότι έγινε ένα πολύ καλό παγκόσμιο φόρουμ το στην όπου είχαμε την ε, δυνατότητα να μιλήσουμε και σε εκπροσώπους από όλο τον κόσμο για το θέμα αυτό. Να σας πω ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ηγηθούμε, θεωρώ, και να προωθήσουμε αυτό το project. Αναμένουμε μια σχετική ανακοίνωση την οποία και θα υποβάλουμε το επόμενο έτος. Να σας πω ότι ένα από τα θέματα τα οποία επί του παρόντος δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλους δείκτες κοινωνικής ευημερίας πέρα από το ΑΕΠ είναι η διαθεσιμότητα, η εγκυρότητα των δικτών αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να ενημερωθεί η διαθεσιμότητα σε ό,τι αφορά τους δείκτες αυτούς και ιδανικά μαζί με την παρουσίαση του ΑΕΠ θα θέλαμε να έχουμε και δείκτες για διαστατικά θέματα. Στην παρούσα όμως φάση δεν έχουμε ακόμα πετύχει κάτι τέτοιο. Θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή και η ανακοίνωση θα, τα... θα εκφράσει αυτό το όραμά μας. για να απαντήσω και στον κύριο Λάμπερτ. Νομίζω ότι απάντησα και στον κύριο Χουντή ταυτόχρονα για το θέμα αυτό του τι γίνεται πέρα από το ΑΕΠ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια των στατιστικών στοιχείων και το ποιος είναι τελικά ο υπεύθυνος. Δημιουργούμε ένα σύστημα όπου η Eurostat έχει ήδη λάβει σημαντικότατες αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά την επαλήθευση upstream των στατιστικών στοιχείων και σε ό,τι αφορά την επιβολή κυρώσεων προς τα κράτη-μέλη για την ε, χειραγώγηση, για την οθεία στατιστικών στοιχείων. Να σας διαβεβαιώσω ότι οι αρμοδιότητες αυτές θα αξιοποιηθούν πλήρως είναι σημαντικό όμως, νομίζω, να μην δοθεί η εντύπωση ότι η τρέχουσα ποιότητα των στατιστικών στοιχείων είναι χαμηλή. Αντιθέτως, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα παράγει πραγματικά στατιστικά στοιχεία υψηλής ποιότητας. Ασφαλώς υπάρχουν προβλήματα γιατί πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο τομέα και αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν. στατ σήμερα έχει σχεδόν όλα τα απαραίτητα μέσα και μέτρα στη διάθεσή της. Σύντομα θα υποβάλουμε μια πρόταση για το ρόλο της Eurostat σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση δικτών για μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες. Και θεωρώ ότι ο κανονισμός αυτός θα δώσει στη Eurostat όλες τις αρμοδιότητες που χρειάζεται για να εξασφαλίσει ότι σε περίπτωση που κάτι κάνουν λάθος τα κρατημέλη στην παρουσίαση των στοιχείων, αυτό δεν θα περάσει σε Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία EGP που παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο, η Eurostat δεν εξέφρασε καμία επιφύλαξη. Αυτό σημαίνει ότι η Eurostat θεωρεί ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για το EDP ήταν αξιόπιστα. Και ότι ακολουθήθηκε όλη η απαραίτητη μεθοδολογία. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Έτζεκ και ο κύριος Σμίτ. Ευχαριστώ. Έχω την αίσθηση ότι αρχίζω και περιμένω με αδημονία τα εισαγωγικά σχόλια του κυρίου Λάμπερτ. Γιατί πάντα κάτι ενδιαφέρον μαθαίνω, είτε για την ειδική του οικογένεια, είτε για τους πρασίνους. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Φιλίπ, λοιπόν, σου λέω ότι μπορεί να έχουν σημασία οι αριθμοί, η ποσότητα, αλλά αυτό που προέχει είναι η ποιότητα. Ο Σβέν Γκίγκολτ και η οικογένειά του είναι καλά. Δεν έχουμε καθημερινή επαφή. Φαντάζομαι ότι είναι με τη γυναίκα και το γιο του αυτή τη στιγμή. Α, εντάξει. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα και συγγνώμη για την προσωπική ε, ερώτηση που έκανα για μια πορεία που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, Θυμάμαι κύριε Επίτροπε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συζήτηση για τις στατιστικές ε, πληροφορίες ε, επ' ευκαιρία της έκθεσης Κλούνα. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κάποια στοιχεία, γιατί εσείς πραγματικά είστε ο αρμόδιος ε, να μας απαντήσετε, γιατί είναι πολύ έγκυρες και οι απόψεις σας. Συζητούσαμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα την ελληνική υπόθεση την ελληνική περίπτωση και ο κύριος Τσικλούνα είπε ότι θα καταρτήσει μια έκθεση που θα μπορούσε να αποφύγει την ελληνική περίπτωση, την περίπτωση δηλαδή που είχαμε με τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία. Κύριε Επίτροπε, ποια είναι η γνώμη σας, τι κλίμα επικρατεί στο Συμβούλιο. Πιστεύετε ότι τα κράτη-μέλη θα είναι πρόθυμα να κοινοποιήσουν σημαντικά στοιχεία για την ευρωπαϊκή μεθοδολογία. Γιατί εγώ αμφιβάλλω μάλλον για την ετοιμότητα ή την προθυμία των κρατών μελών να ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή μεθοδολογία στα θέματα αυτά. Το συζητήσαμε το θέμα εκτενώς την προηγούμενη εβδομάδα και θα ήθελα να ακούσω και τη δική, μας, και τη δική σας γνώμη. Κύριε κύριος Σμιτ. Έχω μία ερώτηση για το φορολογικό θέμα, το, τη δεύτερη αρμοδιότητα του Επιτρόπου. Αφήστε το για το δεύτερο τμήμα. Αργότερα. Αν νόμιζα σήμερα. Ναι, σήμερα, αλλά αργότερα. Είναι το δεύτερο σκέλος της παρουσίασης του Επιτρόπου. Το πρώτο είναι τα στατιστικά, το δεύτερο θα είναι τα φορολογικά. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τον κατάλογο, γιατί παρόλο που δεν ήσταν κύριε Φέη από την αρχή για να ακούσει την παρουσίαση του Επιτρόπου, θα σας δώσω λίγο χρόνο, γιατί δείξαμε μεγαλύτερη πειθαρχία στην τήρηση του χρόνου αυτή τη φορά, οπότε μας έμεινε ε, λίγος χρόνος για τις τελευταίες ερωτήσεις. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ για να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να υποβάλω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις για τα στατιστικά στοιχεία. Η πρώτη ερώτηση αφορά την κατάσταση στη χώρα μου, την Πορτογαλία. Αν η Ευρωστάτ ε, προσθέτει ε, το θέμα, το θέμα της διαχείρισης των, των αεροδρομίων, δεν θα έχουμε πλέον έλλειμμα 5%, αλλά 5,7% γιατί μειώνεται, μειώνονται τα έσοδα και είναι ένα έσοδο που χρησιμοποιείται ε, για να, συνυπολογιστεί στο έλλειμμα. Έχετε εσείς κάποια στοιχεία για το θέμα αυτό, δηλαδή την Πορτογαλία και το θέμα αυτό της ε, διαχείρισης των αεροδρομίων. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει αντίδραση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για παράδειγμα, αν ένα κράτος έχει ένα ευρύτερο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, κάτι που προϋποθέτει ε, σύναψη συμβάσεων. Για κάτι τέτοιο χρειάζονται και εκτάκτο ανάγκης έσοδα και εκτάκτο ανάγκης έξοδα. Έχετε προβλέψει για τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις ε, κάποια μέτρα ή κάποιο τρόπο αντίδρασης. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φέιο, ο Επιτρόπος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Καταρχήν το πρώτο θέμα, το κλίμα που επικρατεί στο Συμβούλιο, την κατάσταση στο Συμβούλιο. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, αύριο το Συμβούλιο θα συζητήσει το στατιστικό πακέτο. Και εξετάζοντας το σχέδιο συμπερασμάτων, ε, θεωρώ ότι αν τελικά φυσικά εγκριθεί αυτό το σχέδιο θα δείξει την ε, στεναρή δέσμευση του Συμβουλίου να προχωρήσει στην έγκριση και να σημειώσει πρόοδο στο κανονισμό. αλλά και ταυτόχρονα να εφαρμόσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών η λογιστικής. Και μια και το Συμβούλιο ήδη κατέληξε συμβαστικές συμφωνίες, τώρα θα πρέπει να οριστικοποιηθούν οι συμβαστικές συμφωνίες μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Πάντως, όταν εγκριθεί αυτό το νομοθετικό πακέτο, φαντάζομαι τα κράτη-μέλη θα κρυθούν να το εφαρμόσουν κιόλα. Και εκεί υπάρχουν δυσκολίες. Πρέπει να εφαρμοστεί και με σωστό τρόπο. Τώρα, για τα συγκεκριμένα θέματα που επισημάνατε της Πορτογαλίας των αεροδρομίων έχω γνώση της κατάστασης και στην επίσκεψη στην Πορτογαλία το επισήμανε και ο υπουργό Οικονομικών της χώρας σας. Αφορά τη διαδικασία EDP για το 2012. Η πρώτη έκθεση θα δημοσιευθεί του χρόνου τον Απρίλιο, γιατί έχουμε και δύο κοινοποίησεις το χρόνο. Θα ήθελα όμως να είμαι σαφής. Όλοι μιλούμε για την ανάγκη της ανεξαρτησίας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και έχουμε και σχέδιο νομοθετικής πρότασης που θα εξασφαλίσει τη δέουσα ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος. Και πιστέψτε με, δεν είναι εναπόκειται στον Επίτροπο σε μένα να αποφασίσει πώς θα χειριστεί την α ή τη β λογιστική πρακτική του, του κράτους, του α β κράτους. Οι, οι στατιστικολόγοι θα εξετάσουν αυτές τις πρακτικές και αυτοί με ανεξάρτητο τρόπο θα λάβουν αποφάσεις, χωρίς καμία όμως επέμβαση ή καμία άσκηση επιρροής από τους πολιτικούς. Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η κατάσταση και αυτό σημαίνει ανεξαρτησία. Και έτσι έρχομαι στην απάντηση στο δεύτερο ερώτημα σας για πιθανές εξαιρέσεις. Δεν θεωρώ ότι με τη θέσπιση των εξαιρέσεων στα στατιστικά στοιχεία μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Αυτό που χρειαζόμαστε στα κράτη-μέλη είναι να εφαρμόσουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι να εφαρμόσουμε τα μέτρα εξυγίανση. Αυτά είναι που θα βελτιώσουν την κατάσταση, όχι εξαιρέσει στη στατιστική διαχείριση της μια μίας ή άλλης δραστηριότητας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και θα περάσουμε στη δεύτερη παρουσίαση για τα φορολογικά θέματα. Και έχω ήδη στον κατάλογο μου πέντε ομιλητές Οπότε παρακαλώ ας δείξουμε επιθαρχή γιατί έχουμε ήδη χάσει 10 λεπτά από την καθυστέρηση της παρουσίασης του Ισπανού Υπουργού. Ελπίζω να μας χορηγήσουν ένα λεπτό επιπλέον οι δερμηνείς. Και παρακαλώ οι ερωτήσεις να είναι σύντομες και να μην ε, σχολιασμοί παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος στην εισήγησή μου και εγώ. Κανείς δεν αμφισβητεί σήμερα πως η φορολόγηση είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της γενικότερης ε, διαδικασίας ε, οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν έχει θέσει επιτάπητος ε, βασικές προτάσεις για να ενισχύσει τη φορολογική διατήρηση, ομοιομορφία στην ενιαία αγορά και να προτείνει χειρισμό των φόρων προς την, με στόχο την ανάπτυξη. Ε, αποταμίευση και ε, φόρος επί των αποταμιεύσεων και φόρος επί των δημοσιονομικών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα πρέπει να σκεφτούμε όχι μόνο ότι είναι ένας παραπάνω φορολογικός φόρτος, αλλά και τη σημαντική συνεισφορά που μπορεί να έχουν αυτοί οι δυο φόροι για την ε, προσπόρωση πόρων. Ε, τώρα, καταρχήν για την αποταμίευση. Πώς μπορεί κανείς να ε, καταστήσει την δύσκολη ήδη κατάσταση της Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιρλανδίας μπλοκάροντας αυτήν την οδηγία. Είναι απαραίτητη και επίγουσα η έγκριση αυτής της πρότασης. Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε γρήγορη πρόοδο σε αυτό το θέμα αναγνωρίζοντας τη σημασία του στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των φορολογικών απατών. Θα ήθελα όλοι οι Υπουργοί Οικονομίας να το θυμούνται αυτό κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο ΕΚΟΦΗΝ αύριο. Στρεφόμενοι στον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, είναι επίση σημαντικό να ταχύτατα να προχωρήσουμε. Ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ισχυρή δημόσια ζήτηση για τον φόρο αυτό, ούτε και τα πολλαπλά ωφέλη που θα μας δώσει από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί. Αφού αποφασίστηκε μετά τις καλοκαιρινές διακοπές ότι δεν μπορούσε να υπάρξει συμφωνία για τον φόρο αυτό σε επίπεδο των 27, λάβαμε επιστολές από 11 κρατημέλη για την έναρξη μια διαδικασία αυξημένη συνεργασία, ενισχυμένη συνεργασία. Το αίτημα διευκρινίζει ότι στόχο και φάσμα αυτή τη πρωτοβουλία θα βασίζεται στην αρχική πρόταση τη Κομισιόν. Προσεκτικά αναλύσαμε το βαθμό στον οποίο αυτά τα αιτήματα συμβαδίζουν με του όρου που προβλέπονται από τη συνθήκη και η απάντηση είναι. θετική ότι, ότι είναι σύμμορφα όλα αυτά με τη συνθήκη. Κατά συνέπεια, έχουμε υποβάλει πρώτα στο Συμβούλιο για να εγκρίνει την ενισχυμένη συνεργασία στον φάκελο αυτό της ε, φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών εφόσον όλα αυτά είναι σύμμορφα με τον νόμο. Η Κομισιόν δεν μπόρεσε να βρει ούτε μία περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ε, συνθήκες, ε, προς τις συνθήκες Πρόκειται για ένα τομέα που καλύπτεται από τη συνθήκη που δεν ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Μετά από εντατικές συζητήσεις δε στο Συμβούλιο, κατέστη σαφέ πως η ενισχυμένη συνεργασία είναι η τελευταία λύση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τώρα, ένα τέτοιο φόρο δεν θα υποβαθμίσει την εσωτερική αγορά. Αντίθετα, θα την ενισχύσει, δημιουργώντα μεγαλύτερη συνοχή και λιγότερο διοικητικό φόρτο για τι επιχειρήσει. Ούτε αυτή η διαδικασία αποτελεί φραγμό στο εμπόριο ανάμεσα στα κράτη-μέλη ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ του. Τέλο, η διαδικασία σέβεται τα δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των μη συμμετεχόντων κρατών μελών. Παραμένουν ελεύθερα να αποφασίσουν και να τροποποιήσουν τη δική του προσέγγιση τη στιγμή που το επιθυμούν. Να μπορούν να αποφασίσουν δηλαδή. Στις επόμενες εβδομάδες το Συμβούλιο θα συζητήσει την απόφαση για να εγκρίνει την ε, ενισχυμένη συνεργασία για τον φόρο δεν θα πρέπει να χάσουμε χρόνο διαδικαστικά για να ξεκινήσει η ουσιαστική συζήτηση. Εγώ από πλευρά μου θα επιταχύνω τη δουλειά τη Κομισιόν για την ουσιαστική πρόταση, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει ανάμεσα στα 11 κατημέλη, ε, αφού θα δοθεί η έγκριση. Μπορώ ήδη να σας επιβεβαιώσω πως η πρόταση αυτή θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αρχική πρόταση της Κομισιόν που εγκρίθηκε πέρυσι. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα σχόλιά σας σήμερα φυσικά θα εξεταστούν πολύ προσεκτικά. Ε, επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το γεγονός ότι ορισμένοι έθεσαν ερωτήματα σε σχέση με τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις ε, του FTT αν αυτό εφαρμοστεί από λιγότερο από 27 χρόνια. Όπως ξέρετε, δε, η Κομισιόν προέβησε εις βάθος ανάλυση για ώστε να στηρίξει την αρχική της πρόταση. Θα αναπτυχθεί περαιτέρω σε επιλεγμένους τομείς που έχουν σημασία στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας, για παράδειγμα για την ενημέρωση των ε, προβλέψεων ε, εσόδων. Ε, θα ήθελα δεν να συγχαρώ την Επιτροπή σας για τη θετική της στάση και για ταχύτητα ταχύτατη εργασία της για το θέμα αυτό. Καταλαβαίνω ότι η Επιτροπή ΕΚΟΝ έκανε ό,τι μπορούσε ώστε να εξασφαλίσει συζήτηση στην Ολομέλεια όσον αφορά τη διαδικασία συγκατάθεσης για την αυξημένη συνεργασία τον Νοέμβριο κιόλα. Σα ευχαριστώ για αυτή την πολύ επικοδομητική συμβολή ε, στην πρόοδο σε αυτό το τομέα και ε, είμαι βέβαιο ότι μπορώ να συνεχίσω να βασίζομαι στην στήριξή σας στα επόμενα βήματα προς μια οριστική εφαρμογή του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Μάλιστα, έχω πολλούς που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις σε αυτό το κομμάτι και εγώ θέλω να θέσω μια ερώτηση και θα το κάνω αυτό γρήγορα γρήγορα ε, μου ζητήθηκε γρήγορα να αντικαταστήσω τον πρόεδρό μας ε, απόψε. Η φοροδιαφυγή, οι απάτες ε, είναι πολύ σημαντικές και ξέρετε ότι οι γαλλικές αρχές ε, έστειλαν στην Google ε, ένα πρόστιμο τεράστιο για βάσματα που έκαναν προς την Ιρλανδία. Και είναι σίγουρο πως ε, πολλές εταιρείες αποφεύγουν ε, να πληρώνουν τους φόρους στα κρατημέλη έχοντας ή μεταφέροντας τις έδρες τους από το ένα κράτο στο άλλο. Δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, γιατί μια μεριά λέτε ότι πρέπει να πείσουμε τους διεθνείς μας εταίρους να συμβαδίσουν μαζί μας και να εφαρμόσουν στους κανόνες, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι εμείς πρέπει πρώτα να βάλουμε τάξη στην Ένωση και να μιλήσουμε για μεγάλη φοροδιαφυγή. Το ίδιο ισχύει και για την Amazon που έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο. Με πολύ μεγάλα θέματα αυτά. Πώς θα το αντιμετωπίσετε, γιατί αυτό είναι εσωτερικό της Ένωσης. Δεν είναι κάποιος διεθνής ε, φόρος ή κάποια μεγάλη φοροαπάτη διεθνού επίπεδου και έπειτα για τον φόρο, φόρο επί των αποταμιεύσεων. Θα ζητήσετε αύριο τα κράτη-μέλη να σα στηρίξουν. Τι κάνετε με το Λουξεμβούργο και την Αυστρία για αυτό το θέμα, γιατί εκείνοι έχουν μια μεταβατική περίοδο. Αλλά και πάλι είναι δύσκολο να πούμε στου διεθνεί μα εταίρου να μα ακολουθήσουν εφόσον δεν συμφώνονται όλα τα κράτη-μέλη τη Ένωση με του κανόνε μα. Ε, τέλος, έχετε άποψη επί αυτών των κρατών που σκοπεύουν να μπλοκάρουν την, αυξημένη, την ενισχυμένη συνεργασία για το FTT επί τη βάση ότι θα στρεβλώσει αυτό την εσωτερική αγορά. Έχετε κάποιο μήνυμα να στείλετε σε αυτά τα κρατημέλη και ποιο θα είναι αυτό. Ας ακούσουμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Κύριε Σμιτ και μετά η κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου κύριε Επίτροπε, αφορά το τελευταίο σχόλιο της ε, κυρίας Μακάρθη για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και τις χώρες που δεν είναι υπέρ. Είχα, διάβασα στην Business Europe μια επιστολή του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου. Φαντάζομαι θα τη διαβάσετε κι εσείς. Εκεί αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι χώρες, ε, οι ευρωπαϊκές χώρες που δεν θέλουν να να εγκρίνουν το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα πρέπει να υποστούν τι αρνητικέ συνέπειες ε, και να αποφευθεί η εξαδαφική φορολογία. Είναι κέριο αυτό το θέμα και ε, επενέσατε την Επιτροπή για την υποστήριξη που σας επιφυλάξε και φυσικά η πλειοψηφία των, επι... των μελών της Επιτροπής είναι υπέρ. Εγώ ανήκω στη μειοψηφία. Μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση τι γίνεται με τις χώρες που θα μείνουν εκτός. Σε ό,τι αφορά το Free CDB, Ακούσαμε τελευταία και Υπουργός Οικονομικών, τον κύριο Όσμπορν, τον κύριο Σόιμπλε, να ζητούν κάποιο είδους συνεργασία σε ό,τι αφορά τον, τον εταιρικό φόρο. Τι γίνεται με το Free πώς έχουν εξελίξεις. Ε, εκεί σας υποστηρίζω αμέριστα, κάτι θα πρέπει να γίνει. Μπορούμε κάτι να πετύχουμε από τους κυρίους Όσμπορν και Σόιμπλε. Κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε και για την πρόταση χρήσης ενισχυμένης συνεργασίας ε, της διαδικασίας αυτής για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για την εφαρμογή αυτής της αρχής, ενώ θα ισχύσει απλή διαβούλευση ως προς την ουσία. Και ε, δεν μου έχει διαφύγει καθόλου αυτή η διαφορά και με ενοχλεί μάλιστα. Δηλαδή η αρχή, η ουσία να διαχωρίζεται από τη διαδικασία. Θα ήταν πολύ καλύτερο και σαφέστερο να μπορούμε να κρίνουμε συγκεκριμένα. Εξηγήστε μου λοιπόν γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκρινε σκόπιμο και χρήσιμο ε, το αίτημά της για την έγκριση του κειμένου για την εφαρμογή του φόρτου χρηματοδοτικών συναλλαγών δεν το επισύναψε. Επίσης, δεν νομίζω ότι είναι πιθανό ο φόρος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών να στηρίζεται στην αρχή της εξοδαφικότητας όπως προβλεπόταν στην πρόταση σας του 2011. Μας είπατε ότι και η νέα πρόταση θα είναι παρόμοια με την προηγούμενη. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, ότι τα κράτη-μέλη που θα θεσπίσουν αυτό το φόρο στο εσωτερικό τους, θα υποχρεώσουν τα, τις χώρες που βρίσκονται εκτός φόρου να εισπράττουν αυτό το φόρο για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που έχουν έδρα στις χώρες που εφαρμόζουν αυτή την ενισχυμένη συνεργασία για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών το κατάλαβα καλά, γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, είναι νομότυπη ε, η νόμη μια τέτοια διαδικασία. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά, γιατί η φορολογική εξοεδαφικότητα θεωρείται ότι μπορεί να επιβληθεί στους υπόλοιπους, ναι ή όχι. Ο κύριος Μπούλμαν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσει έχω να απευθύνω προς τον κύριο Επίτροπο, τον οποίο και ευχαριστώ για την παρουσίασή του. Στη συζήτηση του Six βλέπουμε πάντα ότι και το Συμβούλιο αλλά και η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου έλεγε ότι η προσαρμογή του προπολογισμού δεν ήταν μόνο θέμα ταπανών αλλά και θέμα των ε, εσόδων. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα βέβαια. Η ομάδα μου παρουσίασε μελέτες ε, σύμφωνα με τις οποίες οι αιτήσιες απώλειες, η αιτήσια ζημία ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο φτάνει και το ένα δις ε, απώλειες λόγω φοροδιαφυγής, λόγω κακού συντονισμού, λόγω κακών πρακτικών φορολόγησης. Άρα, λόγω της ύφεση θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Επιτροπές σε μέτα, όταν υποβάλλετε το πρόγραμμα δράσης, δεν θα ήταν καλό να επιταχύναμε κάπως κάποιες νομοθετικές προτάσεις προκειμένου να φροντίσουμε, να φροντίσουμε στην ε, Εαρενή Σύνοδο το Συμβούλιο να λάβει κάποιες αποφάσεις γιατί εμεί θέλουμε να επιταχύνουμε ως κοινοβούλιο, θέλουμε να βάλουμε, να πατήσουμε γκάζι για πολιτική συμφωνία και νομίζω ότι πολλά θα καταφέρναμε να πετύχουμε ε, αν επιτάχυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις διαδικασίες. Ε, κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά το ΕΚΟΦΗΝ και τις συζητήσεις για την οδηγία ε, για την φορολογία. Υποδείξαμε ότι έχει έρθει πια η στιγμή να, κάνουν, να κάνει τις διαπραγματεύσεις ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς ε, οι σοσιαλδημοκράτες το προτείναμε αυτό ήδη το Μάρτιο και δυστυχώς δεν συμφωνήσαν οι συντηρητικοί συνάδελφοι. Αλλά πώς ε, εξηγούν οι Υπουργοί Οικονομικών το γεγονός ότι δεν θέλουν να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν καλούν τους Αμερικανούς να προχωρήσουν σε διεθνή συνεργασία. Αυτό αποτελεί παράδοξο. Πώς το αξιολογείτε εσείς αυτό, Επιτροπές μετά και δεν θα ήταν ε, καλό αν θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τι διαπραγματεύσει εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, λέει η Πρόεδρος. Ε, ελπίζω να μπορέσετε να μα απαντήσετε σε αυτά τα περίπλοκα ερωτήματα. Και μετά θα ακούσουμε κι άλλο ένα γύρο ερωτήσεων. Μάλιστα. Δεν είναι απλέ οι ερωτήσει για τη φορολογία γιατί όλοι είναι εμπειρογνώμονες και ειδικοί σε θέματα φορολογίας. Σε ό,τι αφορά τις δικές σας ερωτήσεις για την φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων και θέματα φοροαπάτης και φοροδιαφυγής γενικότερα. Έχω ήδη ανακοινώσει σε διάφορες περιστάσεις ότι το Δεκέμβριο θα υποβάλουμε ένα πακέτο προτάσεων που θα αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα φοροδιαφυγής και φοροαπάτης. Θα υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις λοιπόν για την αντιμετώπιση των φορολογικών παραδείσων επίσης και των επιθετικών σχεδίων φορολόγησης. Κοιτώντα τα συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία αναφέρατε, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχει ένας, υποθε... ένας επιθετικός προγραμματισμός σε ό,τι αφορά την φορολογία. Θα παρουσιάσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχουν όμως και συγκεκριμένα α, μέσα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ο κώδικας πρακτικών για την φορολογία. Κάθε κάρτος μέλος λοιπόν θα μπορούσε να παρουσιάσει την περίπτωσή του στην ομάδα για τον ε, κώδικα ορθών πρακτικών και εκεί θα αξιολογείται η εκάστοτε κατάσταση από το 97 και μετά έχει προτείνει η ομάδα αυτή να καταργηθούν 100 σχετικές πρακτικές σε κράτη-μέλη. Ύστερα μας ρωτήσατε για το CCTB. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αν εγκριθεί η πρόταση στη CCTB, όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρόβλημα της τιμής, της μεταφοράς τιμών, που συχνά προκαλεί το πρόβλημα της μετάθεσης και μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων σε χώρες με χαμηλότερους μισθούς. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν θα πάψει να υφίσταται στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν προωθούμε την πρόταση για το CCTB τόσο έντερμα. Και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα ασκήσει και ποιήση στο Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο πέρασε η διαδικασία τεχνικής ανάλυσης όλων των άρθρων της πρότασης και τώρα πια έχει έρθει η ώρα να τεθεί στην ατζέντα του ΕΚΟΦΗΝ για πολιτική πλέον συζήτηση. Το έχω συζητήσει με διάφορα κρατημέλη ξέρουμε ότι η επόμενη Προεδρία, πώς να το πω, δεν έχει δείξει ιδιαίτερο ενθουσιασμό για το θέμα αυτό. Αλλά όλες οι Προεδρίες πρέπει να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Άρα, έχει πλέον οριμάσει το, το θέμα, ε, είναι έτοιμο για πολιτική συζήτηση στο ΕΚΟΦΗΝ και νομίζω ότι έχει έρθει πραγματικά το πλήρωμα του χρόνου, να συζητηθούν και τα ωφέλη και σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση ε, επιθετικού προγραμματισμού. Πότε θα τεθεί το θέμα αυτό στην ατζέντα, ρωτάει η πρόεδρο. Δεν είναι ακόμα σαφέ. δεν έχει ξεκαθαρίσει. Αυτό το αποφασίζει η Προεδρία. Το πότε θα μπει στην ατζέντα το θέμα αυτό, η Κυπριακή Προεδρία δεν σκοπεύει να το αναλάβει εξ όσων έχω καταλάβει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, φορολόγηση των αποταμιεύσεων και την τρέχουσα κατάσταση, νομίζω ότι είναι σημαντικό Ξέρετε ότι υπάρχουν... Ε, χρειάζεται ομοφωνία στο θέμα αυτό. 25 κράτη-μέλη υποστηρίζουν ένθερμα την πρότασή μας. Η Αυστρία και το Λουξεμβούργο όμως εξακολουθούν να μπλοκάρουν την πρόταση. Δεν δίνουν καν εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ελβετία. Μπορούμε φυσικά να συζητήσουμε το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, αλλά το να μην δίνει καν εντολή, δυνατότητα διαπραγμάτευση στην Επιτροπή, τι να πω, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και θα το πω μάλιστα ξεκάθαρα στο Συμβούλιο αυτό αύριο. Ελπίζω και οι άλλοι υπουργοί να κάνουν το ίδιο, γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τρεις φορές έχει ζητήσει ποια είναι η πρόοδος για το θέμα αυτό φέτος. Και βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμασταν και πριν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το θέμα τώρα του FTT και της ε, πρότασης. Εν γέννη μάλλον. Κάποιοι μιλήσατε για τα θέματα εξωεδαφικότητας. Κάποια κράτη-μέλη είπαν ότι δεν έχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά αυτό τον εξωεδαφικό χαρακτήρα και ότι η πρόταση η οποία παρουσιάζεται ακολουθεί τις αρχές, τις διεθνείς αρχές και φορολογικές πρακτικές. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η αρχή του κατοίκου που αναφέρεται στην πρόταση προϋποθέτει οικονομικό σύνδεσμο, οικονομική σύνδεση του μέρους που συμμετέχει στην συναλλαγή με το κράτος μέλος που εφαρμόζει τον φόρο και αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί. Μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να αποδείξει ότι δεν υπάρχει τέτοιο σύνδεσμο, τέτοια σύνδεση. Το FCT θα α, μοιάζει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τις πρακτικές που θα εφαρμόζονται με τον ΦΠΑ. Και μπορεί να χρησιμοποιηθούν και τα στοιχεία εξωταφικότητας του ΦΠΑ. Η πρόταση, όπως έχει, δεν έχει οποιοδήποτε αρνητικό αντίκτυπο σε οποιαδήποτε κράτος μέλος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, ενιαία αγορά και τον σχετικό αντίκτυπο, πιστεύουμε και αναφέρεται στην έκθεσή μας αυτό, ότι θα είναι θετικές ε, οι συνέπειες στην ενιαία αγορά. Γιατί αν τελικά επιτευχθεί η συμφωνία μεταξύ των 11 κρατών μελών, αυτό τι θα σημαίνει ότι τουλάχιστον 11 κράτη-μέλη θα έχουν τις ίδιες πρακτικές και τα 16 υπόλοιπα κράτη-μέλη θα έχουν τις δικές τους πρακτικές. Ξέρουμε ότι ο χρηματοοικονομικός τομέας σε διάφορες χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, φορολογείται με διαφορετικό τρόπο και αυτό παρεμποδίζει την αποτελεσματικότητα της ενιαίας αγοράς πραγματικά. Ενώ άμα συντονιστούν τουλάχιστον 11 κράτη-μέλη, αυτό τουλάχιστον θα περιορίσει σημαντικά τον αρνητικό αντίκτυπο. των ενδεχόμενων αποφάσεων των μονομένων κρατών μελών. μην ξεχνάμε ότι Έχουμε ήδη κάποια κράτη-μέλη που έχουν ένα είδος ε, φορολόγηση συναλλαγών και να θυμόμαστε ότι για κάποια μέλη της ομάδας των 11 τα έσοδα από τον φόρο αυτό δηλαδή αν δεν υπάρξει ε, συμφωνία σε επίπεδο των 11 θα εισάγουν το φόρο αυτό μονομερός. Δεν υπάρχει τίποτα που να το εμποδίζει. Και αυτό θα οδηγήσει στη διαμόρφωση ξεχωριστών διαφορετικών πρακτικών. Με μη συντονισμένο τρόπο. Φυσικά, εξετάζοντας τις λεπτομέρειες, διαπιστώνουμε ότι πάντα υπάρχουν διαφορές που τελικά αποβαίνουν ει βάρο του χρηματοοικονομικού τομέα. Μάλιστα, άλλο ένα γύρο ερωτήσεων, η κυρία Ποδηματά και ο κύριο Χοντής και μετά ο κύριο Λάμπερτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την ε, προσήλωσή του στο στόχο της θέσπισης ενός ε, φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών πέραν των σχολείων που κάνατε για την προηγούμενη παρουσίαση και το προηγούμενο θέμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί σεβάστηκε και το γράμμα και το πνεύμα της συνθήκης και προέβησε σαφή διαχωρισμό μεταξύ της ε, έγκρισης ε, της διαδικασίας της ενισχυμένης ενεργασίας ε, από την ουσία αυτής που έχουμε ξεκινήσει ήδη να συζητούμε, αλλά που είναι τελείως διαφορετικό θέμα, διαφορετική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την έγκριση, την σύμφωνη γνώμη δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενισχυμένη συνεργασία, αυτό είναι κάτι που το είχαμε ήδη ζητήσει εμείς. Με την προηγούμενη μας γνωμοδότηση επί της αρχικής σας προτάσεως και είπαμε ρητά ότι αν ε, μία απόφαση σε επίπεδο 27 χωρών μελών δεν καταστεί δυνατή, θα πρέπει παρόλα αυτά να προχωρήσουμε στο μέτρο με τον κανόνα της ενισχυμένης συνεργασίας. Και μετά από εδελεχή εξέταση των ε, σχετικών άρθρων της συνθήκης που αναφέρονται στους όρους ε, εφαρμογής της, του κανόνα της ενισχυμένης συνεργασίας, κρίνουμε ότι πληρούνται πλήρως ε, οι νομικές προϋποθέσεις, οι νομικοί όροι. Εγώ στηρίζω αυτή την πρόταση και αυτό αποφασίσαμε, παραλαμβάνω, ε, επιταχύνοντας και τη διαδικασία. Και μάλιστα πρόκειται να ψηφίσουμε ως όνομα αυτή την πρόταση στις αρχές Δεκεμβρίου, ώστε να επιβεβαιώσουμε την θετική μας στάση και γνώμη ως προς τη διαδικασία της έγκρισης δηλαδή της ε, διαδικασίας της ενισχυμένης συνεργασίας. Τώρα, επί της ουσίας, γιατί πολλά ζητήματα αναφέρθηκαν και πολλά ερωτήματα αναφέρθηκαν στην ουσία. Είπατε ότι εσείς θα εμείνετε πάνω κάτω στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ένας από τους λόγους που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, με μεγάλη πλειοψηφία υποστήριξε την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ήταν το ευρύ πεδίο εφαρμογή της πρότασης που κάλυπτε τα ομόλογα, ε, τα, τις μετοχές και τα εισοδήματα. Θα ήθελα λοιπόν να, ζητήσω επανεπιβεβαίωση εκ μέρους σας με τη νέα πρόταση, αυτή που θα υποβάλλεται μετά την έγκριση της ε, διαδικασίας, της ενισχυμένης συνεργασίας. Θα εμείνετε στο ευρύ πεδίο εφαρμογής που θα καλύπτει ε, μετοχές, ομόλογα και παράγωγα, συγγνώμη, όχι εισοδήματα, παράγωγα και ε, θα λάβετε υπόψη την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βελτιώνει την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί εμείς προτείναμε να συμπεριληφθούν και τα θέματα, το, της, το θέμα της κυριότητας. Σκοπεύετε στην ενημερωμένη σας πρόταση να λάβετε υπόψη και τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και για κάτι άλλο. Επισημάνατε και πάλι την ανάγκη κατεπίγουσας σύνεψης συμφωνίας με την Ελβετία σε ό,τι αφορά τη φορολογία των καταθέσεων. Οφείλω να σας πω ότι εμείς στενιζόμαστε πλήρως τη θέση αυτή, τη γνώμη αυτή και το ίδιο είχαμε πει και πριν από δύο μήνες, αλλά πρώτο δεν βλέπω. Οπότε, τι μπορεί να γίνει ως προς αυτό το σημείο. Επίσης, γνωρίζετε ότι κάποιες χώρες, η πατρίδα μου φέρει πίν, πρόκειται να συνάψουν διμερή συμφωνία με την Ελβετία για την φορολογία καταθέσεων, αποταμιεύσεων. Επειδή θυμάμαι ότι εσείς ήσασταν επικριτικός στη διμερή σύναψη συμφωνίας ε, ε, μεταξύ Γερμανίας και Ελβετίας πριν από δύο μήνες. Πώς βλέπετε αυτές τις διμερείς συμφωνίες. Είστε υπέρ, διάκριστε ευμενός ή θα προτείνατε στις χώρες που προσπαθούν διμερώς ε, να διαπραγματευτούν μια τέτοια συμφωνία να ασκήσουν πιέσεις για πανευρωπαϊκή συμφωνία με την Ελβετία και όχι απλές δημιουργίες. Ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ. Ε, και μένα η ερώτησή μου θα είναι για το φαινόμενο της φοροδιαφυγής από μια άλλη οπτική. Ασφαλώς κύριε Επίτροπε γνωρίζετε ότι υπάρχει πρόσφατη αποκάλυψη της Daily Telegraph για την ύπαρξη μιας νέας λίστας της AGB ε, ε, για τα νησά Τζέρσεϊ όπου περιλαμβάνονται offshore λογαριασμοί. Σε αυτή τη λίστα κατά την εφημερίδα υπάρχουν πελάτες που βαρύνονται με οικονομικά και πολιτικά εγκλήματα, υπάρχουν πελάτες πολίτες μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μου, της Ελλάδας, και ότι αυτή η λίστα βρίσκεται στα χέρια των Βρετανικών αρχών. Αυτή είναι η είδηση. Από εδώ και πέρα αρχίζει η ερώτηση τα στοιχεία αυτής της λίστας όπως και της παλαιότερης λίστας Φαλτσιανή, Φαλτσιάνη, ας με συγχωρέσει ο κύριος που πήρε το όνομα του η λίστα. Στην Ελλάδα αυτή τη λίστα την ονομάζουμε λίστα Λαγκάρντ, διότι η τότε υπουργό Οικονομικών, η κυρία Λαγκάρντ, την παρέδωσε επισήμως στην Ελλάδα. Ρωτώ λοιπόν, τα στοιχεία τέτοιων λιστών, τέτοιων καταστάσεων, μπορούν να διαβιβάζονται νόμιμα μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών. Και το δεύτερο, εφόσον μια χώρα μέλος λαμβάνει τέτοια στοιχεία, μπορεί νομίμως να τα επεξεργάζεται προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες αντιμετώπιση του θέματος της φοροδιαφυγής. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό. Uh, Mr και ο Μάλιστα. Κάθε φορά που σας ακούω, κύριε Επίτροπε, ε, αισθάνομαι ότι είστε όλο και πιο βέβαιος ε, και πιο, με πιο πολύ αυτοπεποίθηση για θέματα φορολογία. και χαίρομαι προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθείτε. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τον ε, φόρο των συναλλαγών, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε η Άννη σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, σε ό,τι αφορά τι αρχέ κτλ. Θα ήθελα να πω δύο λόγια όμως για τα εξωτερικά στοιχεία. Να πω δύο λόγια σε όσους ε, διατείνονται ότι ο φόρος αυτός μπορεί να αποβεί εις βάρος μας. Θα ήθελα ο ίδιος, οι ίδιοι αυτοί συνάδελφοι να μιλάνε για τα ενδεχόμενα, ε, τις ενδεχόμενες βλάβες που θα προκύψουν από άλλες φορολογίες σε κράτη-μέλη. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχουν ως σκοπό να, μειώσουν ε, τους ε, φόρους από τις επιχειρήσεις και ότι έχουμε φορολογικές ιδιαιτερότητες που έχουν ως σκοπό να αυξήσουν ε, τα εισοδήματα από, τον... από τις επιχειρήσεις. Είσαστε κατά των φόρων αυτών. Ας μην ξεγελιόμαστε. Αυτό τι σημαίνει ότι θέλετε να προστατεύσετε τις επιχειρήσεις. Όταν σας ε, εξυπηρετούν τα συμφέροντά σας ε, τα στοιχεία αυτά, τα υποστηρίζετε. Θα πρέπει νομίζω να δείξουμε κάποια ειλικρίνεια. Αυτόφινος, αφετέρου, για το σχέδιο δράσης σας. Αναφέρθηκαν τη διάφορα στοιχεία για το τι θα πρέπει να γίνει ακόμα για την οδηγία για την ε, φορολογία των επιχειρήσεων, των αποταμιεύσεων κτλ. Να πω κάτι για τους φορολογικούς παραδείσους. Ξέρετε ότι έργο ότι το έργο του ΩΣΑ για τους φορολογικούς ε, παραδείσους έχει ξεπεραστεί. εξορισμού δεν υπάρχει προλογική παράδειση και μπορεί κανείς να πάει στο σπίτι του με Ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι ισχύει και ένα θέμα του Μισελ Μπαρνιέ έχει κολλήσει λόγω ξεροκεφαλιάς του. Να σας πω ότι μπορείτε να κάνετε κάτι για να βοηθήσετε το Συμβούλιο να σώσει τα προσχήματα στην ανακοίνωση που προετοιμάζεται στις 4 Δεκεμβρίου. Αν δείξετε αρκετό θάρρος προκειμένου να συμπεριλάβετε μια διατύπωση η οποία θα αποτυπώνει τη θέση του Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά που μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε μια συμφωνία χωρίς ε, να χάσει το κύριο του το Συμβούλιο δεν πιστεύω ότι μας ακούνε και πάρα πολλοί Ευρωπαίοι σήμερα. Ντροπή σε όσους δεν μας παρακολουθούν, τέλο πάντων. Σίγουρα στον τομέα αυτό θα πρέπει να βρεθροποιηθούμε. γιατί ξέρω ότι και εσείς και ο Επιτροπός ε, Μπαρνιέ είστε διδεθειμένοι να κάνετε κάτι για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων, για να μπουν κάποιες βάσεις στο ευρωπαϊκό δίκαιο και να πω ότι πολλά κράτη-μέλη και το δικό μου κράτος μέλος έχουν εντάξει τους φορολογικούς παραδείσους ε, στην ομοθεσία τους για την Ελβετία. Το έχω αναφέρει ήδη. Νομίζω ότι ένα πράγμα μπορείτε να κάνετε και καλύτερα να το κάνει και ο Μπαρόσο, να πάει στην Ελβετία και να της υπενθυμίσει ότι μέχρι το 2014 θα έχουμε επαναπατρίσει όλα μας τα στρατεύματα από το Αφγανιστάν μέχρι τότε θα, έχουν, ε, θα είναι ειδικοί στις ε, ορεινές επιδρομές και τους ξεπερνάμε αριθμητικά. Ίσως αυτό να είναι ένα επιχείρημα. Μπορούμε να ακούσουμε απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις πριν περάσουμε στις επόμενες. Το τελευταίο σχόλιο δεν πρόκειται να το σχολιάσω, να απαντήσω. Δεν χρειάζεται, λέει η Πρόεδρος. Τώρα για τις συγκεκριμένες ερωτήσεις, για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και το πεδίο εφαρμογή στην εμβέλεια της πρότασης και τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως φαίνονται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φαντάζομαι αυτό που θα ακούσετε δεν θα σας εκπλήξει, ούτε θα σας καταπλήξει η πρότασή μας, γιατί ούτως ή άλλως μας δεσμεύουν και οι ε, απόψεις των κρατών μελών που ε, οριοθέτησαν την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη-μέλη έκριναν ότι και η νέα πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να στηρίζεται και να μην απομακρύνεται πολύ από την αρχική τη πρόταση. Δεσμευόμαστε λοιπόν από, τις, από τα αιτήματα των κρατών μελών και δεν μπορούμε να αποκλίνουμε αισθητά από την αρχική πρόταση. Βέβαια θα έχουμε 11 χώρες πια και όχι 27, οπότε θα χρειαστούν κάποιες τεχνικές αλλαγές. Επίσης, εκτιμώντας τους δυνητικούς, το δυνητικ... τις νομικές απαιτήσεις τις νομικές προϋποθέσεις των προτάσεων του Κοινοβουλίου για την συμπερίληψη ε, κάποιων αρχών που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει πρώτα να γίνει η ανάλυση των νομικών επιπτώσεων των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά να δούμε αν θα τις συμπεριλάβουμε. Δεν μπορώ σήμερα να σας παρουσιάσω διεξοδικά την πρόταση. Το καταλαβαίνετε αυτό, αλλά σας διαβεβαιώ ότι δεν πρόκειται η νέα πρόταση να σας ευνηδιάσει, να σας καταπλήξει. Σας καθησυχάζω προς αυτό σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, αποταμιεύσεις και τι μπορούμε να κάνουμε ως προς τη φορολογία τους. Έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση όπου 25 χώρες μέλη δεν θεωρούν ότι χωρούν περαιτέρω παραχωρήσεις ε, προς την Αυστρία και το Λουξεμβούργο. Δεν υπάρχει δυνατότητα να ενδώσουν περαιτέρω στα αιτήματα των δύο αυτών χωρών, οπότε θα χρειαστεί η αναζήτηση πολιτικής συμφωνία ή να ασκηθούν πολιτικές πιέσεις και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς τις δύο αυτέ χώρες για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και τι πρόοδο θα σημειώσουμε. Διαδοχικές προεδρίες πρότειναν πολλές ε, συμβιβαστικές λύσεις στις δύο χώρες αυτές, αλλά απορρίφθηκαν όλες ε, οι συμβαστικές ε, προτάσεις και τώρα έχουμε φτάσει στα άκρα πια, στη... στός εδώ και μη παρέκει. Θα πρέπει όμως να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται, γιατί μερικές φορές ακούγονται και προβάλλονται κάποια επιχειρήματα και στη δημόσια συζήτηση στην Αυστρία και τον Λουξεμβούργο. Όταν μιλούμε για φορολογία των καταθέσεων, των αποταμιεύσεων και ανταλλαγή πληροφοριών, δεν εννοούμε τι καθεστώς θα εφαρμοστεί για τους ε, κατοίκους των χωρών αυτών. Αν δηλαδή η Αυστρία θέλει να κρατήσει το τραπεζικό απόρριτο για του ε, υπηκόου τη, για του κατοίκου τη Αυστρία, του διαβαίνοντε στην Αυστρία, μπορεί κάλλιστα να το κάνει. Αλλά γιατί η Αυστρία να εμποδίζει τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα να φορολογήσει του, τους δικούς της δια, διαμένοντες, τους δικούς κατοίκους με βάση την εθνική της νομοθεσία, τη δική της φορολογική νομοθεσία, γιατί με αυτή την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τους λογαριασμούς αλλοδαπών στη συγκεκριμένη χώρα. Η χώρα αυτή θα μπορέσει να εφαρμόσει τη φορολογική της νομοθεσία με σωστό τρόπο. Γιατί να μπλοκαριστεί αυτή η δυνατότητα, γιατί να αναχαιτιστεί. Κατά τη γνώμη μου δεν ευσταθεί αυτή, αυτό το επιχείρημα. Επίσης βλέπουμε και νέες εξελίξεις παγκοσμίω. Είχαμε τη νέα νομοθεσία στα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, και το Ηνωμένο Βασίλειο, από ό,τι άκουσα ε, για το ΦΑΤΚΑ, έχει υπογράψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, άλλες χώρες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες που κάνουν και τα κρατημέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ως προς τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Καταλήξαμε σε πολύ καλές ε, στερεότυπες συμφωνίες, ε, υποδείγματα ε, συμφωνιών. Έχουμε το πρώτο τέτοιο, τέτοιο υπόδειγμα συμφωνιών μεταξύ, για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κυβερνήσεων και ζητούμε αμοιβαία εφαρμογή. Δηλαδή, εφόσον ε, μια Ευρωπαϊκή κυβέρνηση υποβάλλει, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποβάλλει πληροφορίε προ τι Αμερικανικέ Αρχέ και οι Αμερικανικέ Αρχέ έχουν την υποχρέωση να δίνουν τέτοιε πληροφορίε στη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμε λοιπόν αμοιβαία εφαρμογή, αμοιβαιότητα. Και έχουμε διαπραγματεύσει για να σημειώσουμε πρόοδο. Ό,τι αφορά τι διμερεί συμφωνίε, και εδώ θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρο. αυτό που τα κράτη-μέλη μπορούν να διαπραγματευτούν διμερώς δεν θα πρέπει να εμπίπτει στο, στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Φορολογία Καταθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελβετίας. Τέτοιου είδου θέματα δεν μπορούν να εμπίπτουν σε διμερεί συμφωνίε. Υπάρχουν όμω κάποια θέματα που δεν καλύπτονται από την νομοθεσία για τις καταθέσεις και τη σχετική συμφωνία που θα συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ελβετία. Τέτοιου είδους θέματα που εκπίπτουν τις σχετικές συμφωνίες μπορούν να τα διαπραγματευτούν τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν σαφή όρια λοιπόν. Υπάρχουν θέματα που επιτρέπεται να διαπραγματευτούν τα κράτη-μέλη διμερώς και άλλα που δεν επιτρέπεται. Υπάρχει πάντως το πρόβλημα των καταθέσεων και της συμφωνίας με την Ελβετία. Θα πρέπει να κλείσουμε κάποια παραθυράκια που υπάρχουν και κενά στην οδηγία για τις καταθέσεις και να διαβρύνουμε αυτή τη συμφωνία στην Ελβετία, ώστε η ίση μεταχείριση των καταθέσεων να, να ισχύσει και για την Ελβετία. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Οι διμερείς συμφωνίες δεν παραβλάπτουν ε, ή δεν παρακολύουν το δικό μας έργο για τις ε, καταθέσεις, γιατί το πεδίο εφαρμογή των διμερών συμφωνιών ε, είναι ξεχωριστό από το πεδίο εφαρμογή της σχετικής συμφωνίας που διαπραγματευόμαστε με την Ελβετία. Τώρα για το θέμα των φορολογικών παραδείσων που επισήμανε ο κύριος Λάμπερτ. Ένα από τα στοιχεία που θα προτείνουμε στο πακέτο για τους φορολογικούς παραδείσους θα είναι ο ορισμός τους, ο ορισμός των φορολογικών παραδείσων. Και ευελπιστώ ότι έτσι θα λυθεί και το πρόβλημά σας στις διαπραγματεύσεις που έχετε για την οδηγία για τα κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου. Βέβαια είναι κρίμα που μέχρι τώρα δεν καταλήξαμε σε ορισμό των φορολογικών παραδείσων αλλά πιστεύω ότι με το νέο πακέτο θα καλυφθεί και αυτό το κενό. Τώρα, στην ερώτηση του κυρίου Χουντή για τη λίστα Λαγκάρτ. Και εδώ θα ήθελα να είμαι σαφής. Το θέμα αυτό είναι εσωτερικό. Το, είναι θέμα των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη λαμβάνουν πληροφορίες και εναπόκειται στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν πώς θα αντιμετωπίσουν αυτές τις πληροφορίες, πώς θα τις διαχειριστούν, πώς θα τις επεξεργαστούν και πώς θα εφαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία με σωστό τρόπο. Και δεν θα πρέπει φυσικά να εφαρμόζουν την εσωτερική του νομοθεσία κατά παράβαση των κοινοτικών διατάξεων. Αν διαπιστωθεί τέτοια παράβαση, θα επέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά στο μεταξύ έχουν διακριτική ευχαίρεια τα κράτη-μέλη από τη στιγμή που εθνικά είναι νομότυπες οι παρεμβάσει των κρατών μελών, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρόκειται να επέμβει. Λοιπόν, οι σε σα έδωσαν λίγο χρόνο ακόμη, οπότε μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η κυρία Ρέντινγκ, σύμφωνα με κάποια ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης, είπε σήμερα στο Βερολίνο πως οι ευρωπαϊκές χώρες της Ένωσης δεν θα πρέπει πια να έχουν δικαίωμα άρνηση κυρία σε τόσο λεπτά και αποφασιστικά ζητήματα, καθοριστικά ζητήματα όπως η φορολογία. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσετε τη θέση της κυρίας Ρέντινγκ, αλλά η ερώτησή μου είναι αν είστε της ίδιας άποψης. και ποια είναι η άποψη του υπολείπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το καυτό θέμα. Κέιτ. Ευχαριστώ. Ο Φιλίππο μόλις έφυγε. Αλλά δεν θα ήθελα να πιστεύει ότι τον ηρωνεύομαι για να θεωρήσουμε ότι είναι κάτι το μηδαμινό. Δεν θέλω να το φέρουμε σε αυτό το επίπεδο και να κάνουμε τέτοια σχολεία με την Ελβετή. Θα το, το αναφέρω δημιουργώς. Έχουμε και την ε, ε, οδηγία MIFID όσον αφορά την προστασία του επενδυτή, ιδιαίτερα για τις ε, μικρές επενδύσεις και την ελληνική πώληση. Έχουμε προσταθήσει να προστατέψουμε τους μικρούς επενδυτές. Είναι συχνά οι πιο αθώοι και δεν το λέω αυτό με προσβλητικό τρόπο, αλλά Σίγουρα δεν είναι πολύ πράγμα. Αυτοί που προωθούν τώρα το FTT μέσω ε, της ενισχυμένης συνεργασίας, θα μπορείτε εσείς να τους παρακολουθήσετε πώς ε, θα μετακινηθούν από τους ρυθμισμένους ε, χρηματιστές MIFID και θα παρακολουθήσετε πώς οι μικροί επενδυτές θα προχωρήσουν σε συμβάσεις CFD και την εξάπλωση ε, των ε, στοιχημάτων για τα spreads, γιατί έτσι δεν θα έχουν προστασία όλοι αυτοί. Πολλές από αυτές τις εταιρείε προσφέρουν CFD και στοιχήματα για spreads όπου στρέφονται οι πελάτες μας στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον για τις χώρες όπου σκοπεύουν να εισάγουν αυτόν τον φόρο. Πώς σκοπεύετε να δράσετε. Τελευταίες ερωτήσεις ήταν αυτές. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Σε σχέση με την κεντρική ερώτηση για την ομοφωνία, φυσικά έχουμε την ισχύουσα συνθήκη που μιλάει για ομοφωνία για τα φορολογικά θέματα. Και επίσης έχουμε δυσκολίες όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο. Μόλις σας ανέφερα κάποιες προτάσεις που εδώ και καιρό συζητώνται στο Συμβούλιο. όπου λόγω δηλαδή τη απέτηση τη ομοφωνία δεν μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία. Υπάρχουν κάποιε αρνητικέ πτυχέ τη ομοφωνία. Και φυσικά αυτό καθιστά τη διαδικασία μακρύτερη από όσο θα επιθυμούσαμε. Τώρα, πάντως σήμερα ισχύει η ομοφωνία. Τώρα τι θα είναι αύριο, τι θα γίνει αύριο. Πιστεύω πως θα ξεκινήσουν συζητήσεις για το μέλλον της συνθήκης και αυτό θα είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί. the outcome of, uh, of uh, this debate, but of course taxation is a... Δεν θέλω τώρα να προτρέξω. Φυσικά η φορολόγηση είναι πολύ λεπτό ζήτημα και πρέπει κανείς να, να, να σταθμίσει τα υπέρ και τα κατά πριν να κινηθεί. Επειδή έχουμε ένα πολύ περίπλοκο θέμα που αφορά το FTT και την προστασία των καταναλωτών. Ε, επενδυτών, με συγχωρείτε. Είπατε ότι κάποιοι ήδη προετοιμάζουν ε, σχέδια ώστε να μπορέσουν να παρακάμψουν τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη. Αναφέρεται το Ηνωμένο Βασίλειο Νομίζω πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα έπρεπε να είναι υπέρ της ε, χορήγησης της ε, ενισχυμένης συνεργασίας ε, στα μέλη που το επιθυμούν, διότι αυτό θα μπορούσε να τους ωφελήσει. Αν και δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα συμβεί αυτό. Πάντως, η πρόταση που είναι τώρα επιτάπητος και η νέα πρόταση δεν θα διαφέρει ουσιαστικά από την ισχύουσα, από <coughs> την, ε, μάλλον από την ήδη βληθήσα θα εξασφαλίσουμε ε, ότι θα αντιμετωπίζονται οι δυνατότητες φοροδιαφυγής, θα ελαχιστοποιηθούν και ότι αν χρειαστεί θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν ώστε να ενισχυθούν οι διατάξεις στην πρόταση και να εξασφαλίσουμε πως οι πρακτικές φοροδιαφυγής δεν θα επαληθευτούν. Έτσι λοιπόν πιστεύω θα προχωρήσουμε και αν έχετε κάποια καλή ιδέα για το πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο σχεδιασμό αυτού του φόρου ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ε, φοροαπάτες ή τη φοροδιαφύγη να μας το υποβάλλετε σε μένα ή στους εκπληρογνώμονές μας. Βεβαίω πολλά κράτη-μέλη έχουν ε, επιβάλει τέτοιο φόρο και είναι περισσότερο ακαδημαϊκού επίπεδο αυτή η στους εκπληρογνωμονες μας βεβαιω πολλα κρατη μελη εχουν επιβαλει τετοιο φορο και ειναι περισσοτερο ακαδημαικου επιπεδου αυτη η συζητηση Ναι, ναι, και ήθελα να αναφέρω ότι μόλις ε, ήμουν στην Ινδία και η Ινδία έχει επιβάλει φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών πολύ παρόμοιο, παρεμφερεί με το δικό μας, με τη δική μας πρόταση. Εδώ και αρκετά χρόνια μάλιστα ισχύει. Εφτά νομίζω. Και ρώτησα συγκεκριμένα τον Υπουργό, έχετε πρόβλημα με την ε, με την κατάσταση, φοροδιαφυγή ή αποφυγή καταβολής. Εκείνος όμως με διαβεβαίωσε πως δεν είχαν προβλήματα στην εφαρμογή του φόρου αυτού στην Ινδία. Νομίζω λοιπόν πως όλες αυτές οι ανησυχίες για... με την κατάσταση είναι υπερβολές. Μας περιπτώσει, κλείνει τώρα η συζήτηση γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Επίτροπε, που ήρθατε. Ήσασταν πλήρης στις απαντήσεις σας και Βλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας. Ξέρω πως είναι πολύ δύσκολα όλα αυτά τα θέματα και λεπτά, αλλά όπως είπε και ο κύριος Λάμπερς, είδαμε, σας είδαμε με νέο στένος και ενέργεια και θα μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε. Και ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος, που μας έδωσαν παραπάνω χρόνο, όπως πάντοτε. 13 και 14 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Αύριο δηλαδή, στις 3.